we are going to start the meeting. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση. Χαίρομαι που καλωσορίζω εδώ και πάλι τον κύριο Λελάη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας. Ζητάμε από εσά να μας εξηγήσετε τι έγινε στο Μόντρεαλ. τι έγινε πριν το Μόντρελ και με τις ανησυχίες μας όσον αφορά τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων στις δικές μας ε, δυνατότητες ε, του τομέα του Ευρωπαϊκού Αεροπλοίας δηλαδή. Οπότε είναι σημαντικό να μας εξηγήσετε λιγάκι τι έγινε μετά την συνεδρίαση αυτή και σε λεπτομέρειες πώς θα εφαρμόσουμε το σύστημα αυτό κόρσια ε, και σε σχέση με τα δικαιώματα εμπορίας εκπομπών. Έρχονται και πολλά νέα και από το ΕΚΟΦΗΝ για τη φορολόγηση της κυροζήνης. Οπότε είναι πολύ επίκαιρο το ότι βρίσκεστε εσείς εδώ αυτή τη στιγμή, σε αυτό το πλαίσιο που βρισκόμαστε. Έχουμε και μια νέα επιτροπή, δεν την έχουμε ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει δώσει το πολιτικό της στίγμα για την πράσινη συμφωνία, το Green Deal. Συνεπώς θα σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά και μετά στις πολιτικές ομάδες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι και πάλι εδώ Ανώπων της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος και ευχαριστώ τον ε, Πρόεδρο εδώ που με προσκάλεσε και μου δίνει την ε, δυνατότητα να παρουσιάσω τα αποτελέσματα αυτής της συνέλευσης του ΕΚΑΟ σε ό,τι αφορά το σύστημα της στάθμισης μείωσης εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, στην και ως όταν προσπαθούσαμε να βρούμε ποια θα ήταν η ημερομηνία κατά την οποία θα έκανε αυτή την παρουσίαση. Επιλέξαμε αυτήν εδώ θεωρώντας ότι η νέα επιτροπή θα είχε διοριστεί, θα είχε αναλάβει καθήκοντα και έτσι τα πράγματα θα είχαν ξεκαθαρίσει και περισσότερο. Όμως ε, φυσικά τη σήμερα ημέρα δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν μπορώ και εγώ να προδικάσω το τι ακριβώς θα αποτελέσουν οι πολιτικοί μας ηθήνοντες ε, και η νέα επιτροπή. Μέχρι λοιπόν να διοριστεί και να αναλάβει καθήκοντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές κατευθυντήρε γραμμές, δεν μπορώ να τοποθετηθώ επακριβώς. Επίσης, κατά τελευταία συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ και αναφερθήκαμε σε μια σειρά από ζητήματα, είχα υποσχεθεί ότι θα σας ενημέρωνα σχετικά με, τα, με την, τα όσα συζητούνται στη συνέλευση και το πώς εξελίσσονται εκεί οι συζητήσεις. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό τη υπόσχεση που σας είχα δώσει, βρίσκομαι και πάλι εδώ έτσι ώστε ακριβώς να σας ενημερώσω σε σχέση με αυτές τις συζητήσεις, πράγμα το οποίο φυσικά είναι σημαντικό. Και να σας υπενθυμίσω ότι κατά τελευταία συζήτηση που κάναμε, σας είχαμε αναφέρει εμπιστευτικά και τη θέση της Επιτροπής η οποία συζητήθηκε αργότερα στο επίπεδο του Συμβουλίου και τροποποιήθηκε. Αλλά πράγματι η λόγω συζήτηση έγινε με πολύ αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. Τώρα επιτρέψτε μου να σας πω καταρχήν ότι φυσικά γνωρίζουμε όλοι μας ότι θα πρέπει να μειώσουμε τις ε, κουμπές ε, του άνθρακα και να μειωθεί γενικά η άνθρακα, εκπομπέ άνθρακα ε, στον τομέα τη αεροπορία. Αυτό αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα και η εκλεγή σαν πρόεδρο τη Επιτροπή Φοντρελάνη το έχει θέσει ω μια από τι βασικέ προτεραιότητε. Κατά τελευταία λοιπόν συνέλευση τη ε, ΕΚΑΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει δύο βασικέ προτεραιότητε σε ό,τι αφορά αυτό το σύστημα Κόρσια. Καταρχήν, να διασφαλιστεί μια διεθνή συμφωνία για το Κόρσια και να μην ξεκινήσει και πάλι η όλη η συζήτηση σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που θα συναποτελέσουν το Κόρσια. Και το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι ο στόχος ήταν να διασφαλίσει το χώρο της ε, πολιτικής της ελευθερίας εντός εισαγωγικών, δηλαδή να έχει τα κατάλληλα περιθώρια ευελιξία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρυθμίσει το δικό της σύστημα. Και νομίζω πως ε, στέφθηκαν με επιτυχία και οι δύο αυτοί οι στόχοι μας στο πλαίσιο της ε, συνέλευσης. Καταρχήν θα πρέπει ε, να πούμε ότι πράγματι δεν υπήρξε επαναχώρηση σε σχέση με τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί το 2016, ότι δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο κλαδικό σύστημα για τον τομέα τη πολιτική αεροπορία για τη μείωση των εκπομπών. Ε, στο πλαίσιο λοιπόν αυτή τη συζήτηση με 44 συνολικά χώρε, ε, χρειάστηκε να ταχθούμε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των χωρών εκείνων που θεωρούν ότι το κόρσιο θα πρέπει να είναι πιο αδύναμο ή θα πρέπει να μην περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά του στοιχεία. Εμεί λοιπόν μιλήσαμε με ενιαία φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση παραμέναμε ισχυροί και ταχθήκαμε υπέρ ενός πιο φιλόδοξου συστήματος σε Κόρσια. Και δεν θα είχε διαμορφωθεί με τον τρόπο που διαμορφώθηκε το Κόρσια αν δεν είχαμε ασκήσει πιέσει από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ δεν είναι τέλειο το Κόρσα, Κόρσα και το ανέφερα αυτό κατά τελευταία συζήτηση που είχαμε, αλλά αποτελεί το καλύτερο δυνατό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μα έτσι ώστε να επιτύχουμε παγκόσμιο διεύθυνση σε ό,τι αφορά το περιβάλλον στον τομέα τη αεροπορία, αφού η Συμφωνία των Παρισιών δεν καλύπτει αυτό το τομέα και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των εν στόχων τη Συμφωνία των Παρισιών. Μία δηλαδή παγκόσμια κλίμακα πρόκληση χρήση και μιας παγκόσμιας δέσμευσης και να δράση. Και υπήρξε λοιπόν ε, ε, πλειοψηφία των χωρών που συμμετείχαν στην συνέλευση του ΙΚΑΟ που ε, ψήφισε αυτό το, την πρόταση ψηφίσματο σε αντίθεση με την Κίνα και τη Ρωσία που απέρριπταν ε, το Κόρσια έτσι όπω έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή και ήταν κατά της, του καθορισμού μακροπρόθεσμων στόχων σε ό,τι αφορά τη μίαση των εκπομπών στον αεροπορικό τον τομέα. Είχαμε 92 ψήφους λοιπόν υπέρ και 25 κατά, το οποίο είναι ξεκάθαρο γιατί καταδεικνύει ότι υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία υπέρ του Κόρσια, χωρίς όμως να, αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει ομοφωνία. Καθώς ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να επιτύχουμε την εφαρμογή ε, στο Κόρσια, η υποστήριξη από σημαντική πλειοψηφία ε, χωρών σε οποίε συμπεριλαμβάνονται οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Καναδά, η Ιαπωνία, οι Αφρικανικέ χώρε και οι χώρε του κόλπου, καταδεικνύει λοιπόν ότι ήταν για εμά, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θετικό το αποτέλεσμα αυτή τη ψηφοφορία. Όμω αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε ότι ε, αυτή η διαδικασία κατέδειξε το πόσο εύθραυστη είναι όλη η διαδικασία, του. να επιτύχουμε δηλαδή μια ε, κοινή δέσμευση σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά το κόσμο. Και επίσης ε, ήταν σαφές το πόσο δύσκολο είναι να συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία. Ειδικότερα η Κίνα συμπεριφέρθηκε με τρόπο ε, ή μάλλον συμπεριφέρθηκε ε, σαν να θεωρούσε ότι ήταν απαραίτητη η ομοφωνία προκειμένου να ληφθούν κάποιες ε, αποφάσεις και ε, κατέδειξε επίση απροθυμία να ετηρήσει τι δεσμεύσει τη και τι συνεισφορέ τη. Πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το, ε, τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του συστήματο ΚΟΣΕ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο μα και το τι συνέβη εκεί. Το δεύτερο στόχο ήταν ακριβώ ήταν να διατηρήσουμε, όπω σα είπα, τα περιθώρια ευελιξία στο επίπεδο τη πολιτική μα. Με άλλα λόγια, δηλαδή, ε, εδώ μας ενδιαφέρει ειδικότερα το ζήτημα τη αποκλειστικότητα. Και λοιπόν στο πλαίσιο τη αρχικής συζήτηση, αλλά και στο πλαίσιο των καταληκτικών συζητήσεων και διαδικασιών, δεν ε, έγινε αναφορά στο ζήτημα του, της αποκλειστικότητας ε, του Κόρσια. Άρα λοιπόν δεν αποτέλεσε το αντικείμενο συγκεκριμένη συζήτηση σε αποκλειστικότητα. Έτσι λοιπόν, εμεί με βάση την κοινή θέση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο, δεν χρειάστηκε να θέσουμε κάποια επιφύλαξη σε ό,τι αφορά την πρόταση ψηφίσματος και μάλιστα μια τέτοια ε, ε κίνηση από τη δική μας πλευρά Ενδεχομένω, να, να μείνονται την εντύπωση σε ό,τι αφορά τη δέσμευση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, από τη δική μα πλευρά, από την πλευρά δηλαδή της Προεδρίας, αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο και τη συμφωνία του Σικάγο και των διατάξεων σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση τη ε, κυριαρχία ε, των κρατών μελών ε, και σε ό,τι αφορά και τι υποχρεώσει των συμβαλωμένων μερών σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων τη συμφωνία των Παρισίων, ήταν ξεκάθαρη η θέση μα. και το κάναμε αναφέροντα ότι το μη δεσμευτικό ψήφισμα διατηρεί του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή του να κινηθούμε πέρα ναι, του Κόρσια, ώστε να επιτύχουμε του περιβαλλοντικού μας στόχους σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, εφόσον το επιθυμούμε. Και αυτή η τοποθέτησή μα σημειώθηκε και στα πρακτικά. Επίσης, ε, λόγω σας να υπενθυμίσω ότι αναφέρεται στο ε, δικαίωμα που έχει το, ε, κάθε συμβαλόμενο μέρο να εφαρμόζει την νομοθεσία του στον αεροπορικό τομέα και ασκούμε για παράδειγμα αυτή την, αυτό το δικαίωμα που έχουμε σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφαλεία τη αεροπορία, αλλά και τα περιβαλλοντικά μέτρα τα οποία ήδη εμεί εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ανέκαθεν αποτέλεσε δική μα ε, θέση στο πλαίσιο των ε, διεθνών διαπραγματεύσεων να συνεχίσουμε να έχουμε το δικαίωμα να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά του δικού μα στόχου σε σχέση πάντοτε με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και δεν υπήρξε αντίρρηση στο επίπεδο τη συνέλευση απέναντι σε αυτή τη θέση μα. Οπότε εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να αποφασίσουμε να λάβουμε πιο φιλόδοξα μέτρα εφόσον το επιθυμούμε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα ήθελα να το τονίσω εδώ. Στου επόμενου μήνε τώρα θα εστιάσουμε στην ολοκλήρωση των εργασιών σε ό,τι αφορά το κόστο, ειδικότερα δηλαδή τα offset τη αντισταθμίσεις αν θέλετε, που θα επιτρέψουν ε, την εφαρμογή των ε, κριτηρίων ε, μονάδων εκπομπών. Θα πρέπει δηλαδή να ε, διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει διπλή καταμέτρηση αυτό το double counting δηλαδή σε σχέση με, τα, με τις αντιταθμίσεις ε, το offset και είναι σημαντικό αυτό να το δούμε από κοινού με τη Συμφωνία των Παρισίων στον τομέα δηλαδή της αεροπορίας όταν θα έχουμε καταλήξει και σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 6 της συμφωνία των Παρισίων. Εμείς τώρα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από την πλευρά της Επιτροπής έχουμε ξεκινήσει μια διεξοδική ανάλυση του συστήματος και μόλις θα την ολοκληρώσουμε θα κάνουμε μια παρουσίαση στους συνομοθέτες με βάση και τα όσα προβλέπει και σε συμμόρφωση με την οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS. Ε, και βέβαια θα πρέπει να πω εδώ ότι εμείς παρά τη φιλοδοξία μας δεν μπορούμε από μόνοι μας να ε, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της, των αυξημένων εκπομπών γιατί ε, θα πρέπει όλες οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλο μερίδιο σε αυτές τις εκπομπές να ε, συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια και αφού θεωρείται πως θα αναπτυχθεί περαιτέρω αεροπορικός τομέας ε, αλλού το δικό μας κομμάτι σε ό,τι αφορά αυτές τις εκπομπές θα, θα μειωθεί στο μέλλον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει συμπλήρωση της ευρωπαϊκής δράσης που αναλαμβάνουμε από παγκόσμια δράση. Και από εκεί και μετά, στη συνέχεια αυτή τη παρουσίαση, από το Συμβούλιο θα γίνει μια εξέταση του πώ μπορεί να εφαρμοστεί το ΚΟΡ σε πάντοτε συμμόρφωση με το σύστημα ETS. Επίση, ένα από του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο τη συνέλευση για το Κόρσια ήταν το να δούμε πώ μπορούμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη μείωση των κομπών διοξιδίου του άνθρακα στον ε, διεθνή αεροπορικό τομέα. Και ε, πραγματικά ε, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σα ανακοινώσω ότι καταφέραμε να προχωρήσουμε εδώ γιατί αποτέλεσε άλλωστε και προτεραιότητα τη συνέλευση ηγείων να, δώσει, να, να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και κατά την επόμενη συνέλευση, συνοδευόμενο από έναν οδικό χάρτη, χάρτη πορεία ο οποίο θα εξηγεί το πώ ακριβώς θα επιτευχθεί. Και βέβαια αυτό το ζήτημα θα αποτελέσει προτεραιότητα και για μα για την Επιτροπή και θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα έχουμε στην επόμενη συνέλευση ήδη συγκεκριμένου μακροπρόθεσμου στόχου, αλλά θα έχουμε διασφαλίσει ότι θα έχουν λάβει χώρα όλε οι προπαρασκευαστικέ εργασίε έτσι ώστε να το κάνουμε αργότερο. Και ταυτόχρονα βέβαια η κλιματική διπλωματία θα πρέπει να μα υποστηρίξει στο να πείσουμε όλε τι χώρε να συμφωνήσουμε αυτού του μακροπρόθεσμου ε, στόχου. Δύο λεπτά και ακόμα, Πρόεδρε. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα βιώσιμα καύσιμα στο τομέα τη αεροπορία, εμεί επιέσαμε για ένα πιο φιλόδοξο ε, κείμενο, αλλά δυστυχώ δεν ήταν δυνατό να το επιτύχουμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, το ψήφισμα ε, και η έκκληση που κάνει η συνέλευση ε, αναφέρονται συγκεκριμένα σε πιο βιώσιμα καύσιμα ε, στην αεροπορία. Εμεί θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσει σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε και συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο των φιλόδοξων στόχων της ε, Ένωσης να, μειωθεί, ε, να μειωθούν οι εκπομπές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συγκεκριμένο ποσοστό αντιστοιχεί στο 0,5% σε ό,τι αφορά τη χρήση του ΣΑΠΣΑ και αυτό οφείλεται βέβαια και στην έλλειψη των υποδομών, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει στο μέλλον μια σημαντική συνεισφορά. Όμω θα πρέπει να υπάρξει ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να δώσει τα απαραίτητα κίνητρα για τι επενδύσει, για την καινοτομία εδώ έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε ακριβώς τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και την υποκατάσταση της κυροζήνης. Τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάποιε συγκεκριμένε δεσμεύσει ε, σε, ό,τι αφορά την ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σίγουρα είμαστε υπέρ ε, της τη ε, υποστήριξη των εναλλακτικών καυσίμων και τη εμπορευσιμότητά του. Δηλαδή, του να είναι σε θέση πλέον να, να είναι βιώσιμα δηλαδή, αυτά τα καύσιμα οικονομικά. Επίσης, ο στόχος μας προφανώς είναι έχουμε σημαντική μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 5% και ε, για να το επιτύχουμε αυτό θα χρειαστούμε φυσικά ε, ένα πλήρες, μια πλήρη δέσμη, αν θέλετε, μέτρων, ένα συνδυασμό μέτρων ε, στα οποία συγκαταλέγεται ακριβώ και η εφαρμογή του συστήματο Κόρσια. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να δούμε και άλλα στοιχεία, όπω για παράδειγμα οι, ε, οι ενισχύσεις και οι φοροαπαλλαγές που δίνονται στις ε, αεροπορικές εταιρείες. Επίσης, εκείνο που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι και το σύστημα ΣΕΖΑΡ και ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, έτσι ώστε δηλαδή να κάνουμε τις αντίστοιχες προσπάθειες και ήδη έχουμε εξοικονομήσει 2,6 τόνους ε, διοξιδίου του άνθρακα από το 2015 και θα μπορούσαμε με τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό ε, να επιτύχουμε ακόμα περισσότερο εφόσον βέβαια σταματήσουν να μπλοκάρουν αυτή την πρωτοβουλία τα κράτη-μέλη όπως το κάνουν εδώ και χρόνια. Άρα λοιπόν ε, Πρόεδρο, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να φτάσουμε σε μια πραγματική φιλοπεριβαλλοντική αεροπορία αλλά αυτός παραμένει ο δικός μας στόχος και θα εντατοκοποιήσουμε τις προσπάθειές μας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι ώστε να φτάσουμε σε αεροπορικέ μεταφορέ με μηδενικέ εκπομπέ. Και φυσικά εδώ βασιζόμαστε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναμένω με ενδιαφέρον τα ερωτήματά σα και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και για το παραπάνω χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστούμε. ερωτήσει τώρα. Πίτερ Λίζα, ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ τον Γενικό Διευθυντή. Θέλω να αρχίσω με δύο σημεία με τα οποία συμφωνώ μαζί σας. Πρώτα απ' όλα για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Πράγματι, είναι ένα θέμα που πρέπει να πετύχουμε. Και επί όταν ε, μιλάτε για καύσιμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, οποιοδήποτε μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αποτελεί μέρος του πολιτικού μείγματος, όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς. Αλλά για τα καύσιμα αυτά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα ε, στην οδηγία ε, για τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας μπορεί να κάνει περισσότερα για την αεροπορία. Δεν νομίζω ότι κάνει αρκετά. Όσον αφορά το Κόρσια τώρα, το σύστημα Κόρσια, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε ευτυχείς. Και δεν είναι αυτή η θέση της Επιτροπής ένβη μόνο, αλλά ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμεί δεν πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη καμπή εδώ. Έχει πολλά κενά, είναι πολύ αδύναμο αυτό το σύστημα και δεν ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία των Παρισίων, ούτε με τα όσα μας ζητάει η επιστήμη να κάνουμε. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας λόγος για να εκφράσουμε το θυμό μας και απέναντι στους υπουργούς μεταφοράς και απέναντι στην ΜΟΥΒ, γιατί τελικά έχουμε την αίσθηση ότι δεν πρόκειται για υπουργού μεταφοράς, αλλά υπουργού αεροπορίας. Αυτό που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ευνοούμε την αεροπορία με λιγότερη φορολογία, ε, με λιγότερες φιλοδοξίες στο ETS και οι συνόδρομοι φορολογούνται υψηλότερα μα Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο πια. Είχαμε αυτή την στάση για πολλά χρόνια και τώρα είναι προτεραιότητα για τους εκλογείς μας να αλλάξει αυτό. Το σύστημα Κόρσια λοιπόν δεν φτάνει για να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό και την επιθυμία των πολιτών. Και τώρα έρχομαι στο πολιτικό ζήτημα της συναπόφασης. Και εδώ θέλω πραγματικά να σας ζητήσω να επιβεβαιώσετε ότι όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές στο τραπέζι και μόνο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν το τι θα γίνει με το σύστημα δικαιωμάτων εκπομπών. Φυσικά και μπορούμε να αυξήσουμε τη φιλοδοξία, μπορούμε να πάμε σε ένα πλήρη πληστηριασμό. Και η κυρία Φοντερλάιν προς αυτή την κατεύθυνση πάει, όχι βήμα-βήμα, αλλά πλήρης πληστηριασμός. Και επίσης να το έχουμε για τις διπυρωτικές πτήσεις το ETS. Αυτό πρέπει να είναι μία επιλογή. Ερμηνεύετε κι εσείς έτσι τα πράγματα. Και αν όχι, γιατί έχετε παρετηθεί από αυτό το προνόμιο του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Θα ακούσουμε πρώτα τις ερωτήσεις των συντονιστών, θα τις απαντήσετε και μετά θα περάσουμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Λοιπόν, έχουμε ήδη δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις από τον Πίτερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Γκέτλαντ. Ε, σας ευχαριστώ, Γενική Διευθυντά, που ήρθατε εδώ. Έχετε ξανάρθει και χαίρομαι γι' αυτό. Για τους σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί μείωση των εκπομπών από ολόκληρη την κοινωνία και κυρίως από τους κλάδους αυτούς που εκπέμπουν περισσότερο όπως είναι η διεθνής αεροπορία. Και η ιδέα πίσω από το σύστημα Κορσία δεν είναι κακή. Έχει νόημα να έχουμε ένα συνολικό πρόγραμμα για ένα συνολικό ε, πρόβλημα. Έχετε ξανάρθει εδώ, όπως είπα, οπότε γνωρίζετε ότι η Επιτροπή μας έχει εκφράσει ε, και παλιότερα πάρα πολλές ανησυχίες όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος αυτού. Έχω βέβαια λιγότερα ερωτηματικά όσον αφορά την Γενική Συνέλευση και το σύστημα Κόρσια, αλλά θα έρθω σε αυτά που θα σα ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα το θέμα της αποκλειστικότητας. Άρθρο 18 λέει με σαφήνεια ότι το σύστημα Κόρσια είναι το μόνο διεθνές μέτρο που αναφέρεται ε, στις περιορισμούς των εκπομπών σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το Συμβούλιο τώρα και η Επιτροπή λένε ότι δεν είναι πρόβλημα αυτό και ότι δεν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αμφισβητήσει αυτή τη διατύπωση. Γιατί εγώ δεν είμαι πεπισμένη. Ε, πώς καταλήξατε νομικά σε αυτό το συμπέρασμα. Και μια που συζητάμε θέματα που έχουν να κάνουν με το σύστημα ETS, να πούμε κάτι άλλο. Το άρθρο 30 στην οδηγία ETS ε ρητά υποχρώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει πώς θα λάβει υπόψη μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 ότι δεν έχει να κάνει με το εκπομπέ οξυδιού του άνθρακα. Οπότε θέλω να ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανταποκριθεί στην προθεσμία αυτή. Και δεύτερον, πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την έκθεση αντικτύπου για να διασφαλίσει ότι όλες οι υποστημονικές απόψεις αντικατοπτρίζονται στη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ρινιού. Ναι, σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορώ να πω εδώ πέρα περισσότερο όσον αφορά την διατύπωση αυτή. Τα είπαμε και στις 4 Σεπτεμβρίου. Εσείς μιλήσατε για silver bullet και το είπατε και το ξανάπατε. Και εξηγήσατε με ποιο τρόπο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι συγκεκριμένα μέτρα Κανενός είδου μέταλλο δεν θα μας έκανε. Δεν είναι μόνο το ασίμι που μας ενοχλεί στο Silver Bullet. Τώρα, είναι ένας τρόπος για να αποφύγουμε βασικά το θέμα. Είτε πρόκειται για διανοητική βαρεμάρα, είτε πρόκειται για πολιτική ανικανότητα. Και θα έπρεπε να είσαστε σε θέση να δείτε όλες αυτές τις ε, αποφάσεις. Δεν είναι θέμα να μας παρουσιάζεται έναν ρόδινο πίνακα ότι όλα είναι καλά και δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Και αν εσείς δεν το βλέπετε αυτό, τι να πω. Δεν θα αποκτήσετε πολλούς φίλους στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Πράσινη τώρα, ο Μπάς. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ τον κύριο Λαλάη. Ε, νομίζω ότι επαναλαμβανόμαστε εδώ. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι θλιβερό, δεν είναι. Οι επικρίσεις παραμένουν. Και εσείς δείχνετε να υποστηρίζετε ότι ό,τι συμβαίνει στο διεθνές επίπεδο είναι καλό. Εγώ δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο. Και πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, πιο επικριτικοί, δεδομένου ότι επίγει να περιορίσουμε τις εκπομπές μας και κυρίως αυτές της αεροπορίας. Και εδώ ήδη το ότι επίγει το θέμα είναι το σημαντικό και όταν σας ακούμε δεν το βλέπουμε αυτό. Ακούγεται σαν, ακούγεστε σαν εκπροσωπείτε την ΙΚΑΟ και μην το παίρνετε θετικά αυτό, δεν το λέω για καλό. Λοιπόν, δεν θέλω βέβαια να πάω πολύ πίσω, αλλά να ξέρετε ότι εγώ ε, δυσκολεύομαι. Το Σεπτέμβριο συζητήσαμε το κατά πόσο θα έχουμε επιφύλαξη όχι, εσείς συζητήσατε στο Συμβούλιο. Αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υπέρ της επιφύλαξης, στο Συμβούλιο όμως είπε όχι, ας αποφασίσουμε στο Μόντρεαλ. Και τώρα έρχεστε και λέτε, μα δεν ήταν θέμα συζήτησης, ωραία δεν ήτανε. Μα τι λέτε τώρα. Τι έγινε με την αρχική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς θέλατε την επιφύλαξη. Δεν έχει αλλάξει το κείμενο στο μεταξύ. Οπότε τι είναι αυτό που άλλαξε και τώρα δεν θέλετε την επιφύλαξη και λέτε ήταν πολύ καλό το ότι δεν έγινε συζήτηση γι' αυτό και άρα δεν χρειάζεται να υποβάλλετε επιφύλαξη. Εδώ μας, μας φαίνεται σαν να προσπαθείτε να κάνετε τα χατήρια του ΙΚΑΟ και ξεχνάτε τις αρχικές ανησυχίες που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι θέλουμε να υποβάλουμε την επιφύλαξη. Εδώ δεν βλέπω συνέπεια από την πλευρά σας, αλλά σκετάξουμε κοιτάξουμε και λίγο προς το μέλλον. Λέτε ότι δεν μπορείτε να πείτε τα πάντα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό όμω που ξέρουμε είναι ότι η American Airlines σας γράφει για τι φορολογικές γερμανικές πρωτοβουλίε και λένε ότι η Κορσία πρέπει να παρεύει και ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίε είναι σε βάρος της Κορσίας. Μα αυτό σας δείχνει πώς χρησιμοποιούν ε, Πώ χρησιμοποιεί ο κλάδο την κορσία. Αυτό δεν θα έπρεπε να σα ανησυχεί. Δεν θα έπρεπε αμέσω να του απαντήσετε και να του λέτε σταματήστε. Δεν πρόκειται και ω Ευρώπη θα αναλάβουμε τι δικέ μα ευθύνε. Γιατί εσεί λέτε ότι ίσω μπορεί να μην υπάρξει διαμάχη νομικά. Ξέρετε όμω ότι πολιτικά θα τη χρησιμοποιήσουν την κορσία και τη χρησιμοποιούν οι ίδιοι American Airlines. Τι θα κάνετε λοιπόν γι' αυτό. Και τέλο. αυτά που ρώτησαν κι άλλοι. Τον Ιανουάριο το 2020 θα έρθει η Επιτροπή με μία έκθεση για, για την ρήπανση. Εσείς τι θα κάνετε, θα είσαστε έτοιμος να δράσετε τότε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ομιλητής ε, συντονιστής από το ID, το ECR. Ο Αλεγάνδη Φωτρά, όχι. Από την ΚΟΕ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέτε ότι το καλύτερο διαθέσιμο μέσο είναι το Κορσία. Είπατε ότι είναι το καλύτερο διαθέσιμο. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάποιο καλύτερο το οποίο να διαθέτουμε, αν όντω ισχύει αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πάρα πολλά ελαττώματα και πρέπει να το καταργήσουμε. Χρειαζόμαστε να αντικαταστήσουμε τις προσεγγίσεις ε, της αγοράς με ε, ε, αποτελεσματικά δεσμευτικά ρυθμιστικά συστήματα. Η εμπορία εκπομπών και τη διάθεση στην αγορά είναι χειρότερο από το να μην κάνουμε τίποτα. Είναι παραπλανητικό και πολλοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι σίγουρα συμβάλλει σε καθαρή αύξηση στο ε, απόλυτο ποσοστό των εκπομπών. Από το 2020 οι παγκόσμιες εκπομπές θα είναι περίπου 70% υψηλότερες ε, στην αεροπορία από ό,τι τώρα και αναμένεται να αυξηθούν πάνω από 300% μέχρι το 2050. Ο ΙΚΑΟ ε, φαίνεται ότι δεν έχει κάποιο σχέδιο για να μειώσει αυτή την αύξηση λέει ότι θέλει να έχει ε, ουδέτερος προς τον άνθρακα ε, καύσιμα, να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά καύσιμα κλπ. Αυτό είναι παράλογο. Ε, είναι σαν να αντικαθιστάτε τα καύσιμα με βιοκαύσιμα. Τα πιο φθηνά διαθέσιμα βιοκαύσιμα για την αεροπορία ε, παρασκευάζονται από συγκεκριμένε εταιρείε οι οποίε οδηγούν σε τεράστια αποψήλωση των δασών. Χάνουμε λοιπόν και από τι δύο πλευρέ δεν υπάρχουν διαθέσιμες ε, λύσεις ε, για τον τομέα της αεροπορίας για να σταματήσει να καίει ορυκτά καύσιμα αυτή τη στιγμή. Μήπως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συχνές πτήσεις ε, και να σταματήσουμε να επεκτείνουμε τα αεροδρόμια. Η αένα η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή και δεν είναι βιώσιμη σε έναν πλανήτη ο οποίος είναι πεπερασμένος και η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία είναι μια αποτυχημένη ιδεολογία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε αυτό ο πρώτος γύρος πολύ συγκεκριμένων ερωτήσεων και περιμένουμε συγκεκριμένε απαντήσεις από εσά. Σας ευχαριστώ και προσπαθήστε να είστε συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Και φυσικά και για τις επικριτικές ερωτήσεις, διότι και αυτές είναι σκέλος ε, της συζήτησης που κάνουμε. Και ε, συμμερίζομαι και εγώ την αίσθηση του κατεπήγοντος εδώ και συμφωνώ ότι σίγουρα το Κορσία δεν είναι η ιδανική λύση, αλλά και πάλι πρέπει να πω ότι είναι η μόνη παγκόσμια λύση και αυτό το οποίο και εμείς επιθυμούμε να δούμε είναι να υπάρχει πολυμερής δέσμευση με τους εταίρους μας. Πρόκειται για ένα πολυμερές βήμα λοιπόν και τα πολυμερή βήματα σημαίνουν και δυστυχώς συμβιβασμούς προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ε, ε, που θα συμμετέχουν. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Και βεβαίως αυτό είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η παγκόσμια πρόκληση στην αεροπορία, γιατί θέλουμε και οι άλλες περιοχές να δεσμευτούν και να θεσμευτούν σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Τώρα, θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε μια σειρά από παρατηρήσεις που έγιναν, ξεκινώντας με την ίδια σειρά με τον Πίτερ Λίζε όσον αφορά τα καύσιμα τα οποία είναι ουδέτερα ω προς τη χρήση του άνθρακα. Συμφωνώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και σας εγγυώμαι ότι πλέον εξετάζουμε πάρα πολύ σοβαρά αυτή την περίπτωση και προσπαθούμε να βρούμε μια σωστή λύση η οποία θα λάβει υπόψη ε, επίσης ε, και σημείωσα και τις παρατηρήσεις ε, για τα βιώσιμα καύσιμα τα οποία μπορεί να έχουν ε, αρνητικό αντίκτυπο στην αεροπορία. Ε, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οτιδήποτε θα επιλέξουμε πρέπει να το λάβουμε υπόψη και νομίζω ότι εδώ ό,τι κάνουμε ήδη μας βοηθά να προχωρήσουμε. Σημείωσα επίσης και τις επικριτικές παρατηρήσεις σας για το Κορσία ε, δεν με εκπλήσει. Ξέρω ότι πάντα ζητούσατε πολύ περισσότερα από όσα ε, έχουν ε, γίνουν δεκτά, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει δέσμευση σε αυτή τη διεθνή διαδικασία. Χωρί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρί την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η διεθνή προσέγγιση κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχε οδηγήσει πουθενά. Και τώρα θα είχαμε ακόμα μια κατάσταση ε, μάλλον έχουμε 81 χώρε οι οποίε συμμετέχουν εθελοντικά και είναι το 66% τη διεθνή αεροπορική δραστηριότητα. και υπάρχουν 91 χώρε οι οποίε είναι υπέρ του Κορσία. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει παγκόσμια δέσμευση την οποία δεν θα είχαμε καταφέρει με άλλο τρόπο και εδώ προσπαθούμε συνεχώ ε, στι τεχνικέ συζητήσει να αυξήσουμε την ακαιρεότητα του Κορσία. Δεν έχουμε μείνει αδρανεί. σα ίσα η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και πιστεύουμε ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε και αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα τα θέματα της φορολόγησης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό είναι τμήμα αυτών των συζητήσεων που βρίσκονται επιτάπητος Και σίγουρα θα θέλαμε και τα άλλα μέσα μεταφοράς ε, να προτείνουν βιώσιμες ε, λύσεις ε, και δεν λέω μόνο ότι εδώ κολακεύουμε και μόνο. Υπάρχει και η Connecting Europe Facility και περίπου το 75% ε, δόθηκε για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών συστημάτων και επίσης στις εσωτερικές πλωτές οδούς που είναι ένας ε, περιβολοντικά φιλικός ε, τρόπος μεταφοράς και το 90% που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δοθεί για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Όσον αφορά το μέλλον της φορολογίας, αυτά είναι ένα από τα θέματα τα οποία βρίσκεται επιτάπητος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας είπαν ότι εξετάζουν για την οδηγία για την ενέργεια και την ενεργειακή φορολόγηση. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις που έχουν ε, ξεκινήσει ε, να συζητούνται και σε διάφορες συνθέσεις, ε, ήδη και στο ΕΚΟΦΕΝ, ε, στο ΕΚΟΦΗΝ ε, θα φτάσουν κάπου και οι πολιτικοί φύνοντε θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις. Επομένως, ε, οι συζητήσει αυτές είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τις επιλογές, ναι, βεβαίως, οι επιλογές όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορία της Εκπομπών υπάρχουν. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν έχει απορριφθεί και θα τις εξετάσουμε όλες. Δεν θέλω βεβαίως να προδικάσω το αποτέλεσμα της μελλοντική Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε τη δέσμευσή μας με το Κορσία με την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάμε πέραν του Κορσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες. Και νομίζω ότι αυτό ε, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση και θα μας επιτρέψει να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε και το χώρο πολιτικής μας. Το είπα προηγουμένως και θα συνεχίσω να το λέω. Έχουμε διατηρήσει το χώρο πολιτικής μας. Εμείς μπορούμε να λάβουμε τις αποφάσεις μας ε, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούμε να εφαρμοστεί αυτό στην Ευρώπη, σε αυτή την περιοχή και αυτό ε, συνάδει πλήρως και με τη σύμβαση του Σικάγο. Υπήρχε και ένα θέμα όσον αφορά τη συνέπεια της Κορσία με τη Συμφωνία του Παρισιού και την ε, ανάπτυξη του 2020 που συμφωνήθηκε από τη συνέλευση και είναι το πρώτο βήμα για τη μείωση των εκπομπών της αεροπορίας. Ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω βελτιωμένης τεχνολογίας αεροσκαφών, τεχνολογικών βελτιώσεων, εισαγωγή βιώσιμων καυσίμων στην αεροπορία, αλλά και συγκεκριμένων μηχανισμών της αγοράς ε, του συστήματος εμπορίας εκπομπών και του Κορσία. Ε, είναι οι τέσσερις ε, κλάδοι στους οποίους θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και τα αποτελέσματα σε όλα αυτά τα παρακλάδια προκειμένου να μπορέσουμε να μειώσουμε και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της αεροπορίας. Το Κορσία καλύπτει πολλές χώρες όπως είπα και αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες και φυσικά αφορά και αερογραμμέ οι οποίες ε, ε, πετούν σε διαδρομές μεταξύ αυτών των χωρών. Τώρα, όσον αφορά την αποκλειστικότητα, και νομίζω ότι εδώ είχαμε αρκετούς συντονιστέ ε, που έφυξαν αυτό το θέμα. Ναι, το συζητήσαμε εδώ. Ενομερωθήκατε και για τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν πάμε στη συνέλευση της ΑΙΚΑΟ. Αλλά ταυτόχρονα η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ε, και η θέση αυτή τροποποιούσε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και αυτό φυσικά είναι δικαίωμα του Συμβουλίου να αποφασίσει τη θέση της Ένωσης βάσει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως η προφορική δήλωση που έκανε η Προεδρία εκ μέρους του Συμβουλίου εξασφαλίζει ότι και πάλι θα διατηρήσουμε το χώρο πολιτική μας και θα εγγυηθούμε και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά δεν δρούμε κενό στις ε, διεθνείς διαπραγματεύσεις. Πρέπει να βασιζόμαστε και εντός του πλαισίου που παρέχεται και σε αυτή την περίπτωση με τη θέση της Ένωσης και η θέση της Ένωσης καθορίζεται από τα κράτη-μέλη όπως ε, έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Και βάσει της συμφωνημένης ευρωπαϊκής θέσης η συνέλευση αξιολόγησε την κατάσταση επιτόπου για να μπορέσει να προφυλάξει το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και το χώρο Πολιτική και κατέληξε ότι σε καμία από τι κόκκινε γραμμέ που είχαμε καθορίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχε πρόβλημα. Δεν ε, ξεπεράσαμε καμία από αυτέ τι γραμμέ. και φυσικά η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και τα ε, κράτη-μέλη της ΆΙΚΑΤ πήραν το λόγο και πίεσαν συνεχώς για την αποτελεσματικότητα του Κορσία και φυσικά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Όπως σας είπα και προηγουμένως, το ψήφισμα της συνέλευσης του ΑΕΚΑΟ δεν είναι νομικά δεσμευτικό και σε καμία περίπτωση δεν απαιτεί συμμόρφωση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομοθεσίας των κρατών μελών. Αυτό το ψήφισμα ε, αναφέρεται και στην αποκλειστικότητα για ένα παγκόσμιο σύστημα. Το ευρωπαϊκό σύστημα είναι περιφερειακό. Επίσης, ε, βάσει και της ε, σύμβασης του Σικάγο, κάθε συμβαλόμενο μέρος μπορεί να εφαρμόσει ε, χωρίς διάκριση την ε, εθνική του νομοθεσία εντός της ε, επικράτειάς του και της δικαιοδοσίας του και αυτό ισχύει και για το δίκαιο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Να επισημάνω λοιπόν και πάλι ότι ο χώρος πολιτικής μας έχει προφυλαχθεί καταλήλως σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα. Just see, uh, Yes, uh, there um, uh, the, question about the, Υπήρχε και μία ερώτηση για τις επιπτώσεις που δεν αφορούν το διοξίδιο του άνθρακα στην αεροπορία, διότι στις πτήσεις έχουμε και ε, θιούχες ε, εκπομπές που έχουν ε, περίπλοκες συνέπειες ε, για την ατμοσφαιρική ρήπανση και είναι γνωστές αυτή τη στιγμή οι γνώσεις που έχουμε είναι από μέτριες έως σχετικά χαμηλές ε, και η οδηγία ε, προβλέπει αντίκτυπο ε, και μελέτη αντικτύπου για τα θέματα αυτά και αυτό έχει ξεκινήσει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αναμένεται του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, αλλά είναι κάτι το οποίο έχουμε στα σκαριά και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε μόλις ε, μπορέσουμε. Ε, ξέρω ότι δεν είναι ιδεώδες ε, να έχουμε καθυστερήσεις, αλλά οι καθυστερήσεις συμβαίνουν και φυσικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διορθώσουμε την κατάσταση και να την αντιμετωπίσουμε. Είχαμε και μία ερώτηση και σχόλια από τον κύριο Τόρβαλτς. Ε, ευχαριστώ και για το εστονικό, ε, την εστονική παράτηση. Θα μπορούσα να απαντήσω στα φιλανδικά, αλλά αργότερα στους διαδρόμους. Τώρα, ε, τίθεται ο προβληματισμός ε, στο ΕΝΙΚΑΟ. Ναι, φυσικά τίθεται συνεχώς και το συζητούμε και σε τριμερές επίπεδο στις διμερείς μας συζητήσεις ε, ε, με τις χώρες αυτές στο περιθώριο αυτών των συναντήσεων. Και πρέπει να πω ότι είναι πολυμερές αυτό το βήμα και έχουμε 193 χώρες οι οποίες έρχονται και από διαφορετικό ε, πλαίσιο και επομένω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, μέγιστη δυνατή πλειοψηφία. Δεν ήταν καθόλου εύκολε οι διαπραγματεύσει και σα εγγυώμαι και επίση μπορώ να σα πω ότι ιδιαίτερα όταν η κινέζικη αντιπροσωπεία πήρε το λόγο ε, ήταν πολύ κρίσιμη η στιγμή. Βλέπετε ότι ήταν σαν να πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο. Είχαμε μπει σε μια μηχανή του χρόνου και πήγαμε στο παρελθόν διότι όλε αυτέ οι συζητήσει είχαν ξαναγίνει. Δυστυχώ. Ε, ξανακάνουμε όμως αυτές τις συζητήσεις. Επομένως δεν υπάρχει διεθνή συνένεση. Η δική μας δουλειά είναι να εγγυηθούμε ότι θα έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους διεθνούς εταίρους να συμμετέχουν και φυσικά ε, και πριν από πέντε χρόνια κάποιοι έλεγαν ότι το Κορσία θα είναι καταπληκτικό και μόλις... Ε, ε, συσταθεί και αρχίσει να έχει πραγματική περιβαλλοντική ακαιρεότητα, θα αρχίσει να αλλάζει τα πράγματα γιατί είναι παγκόσμιο και συμμετέχουν όλοι. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι προσδοκίε είναι πολύ μεγαλύτερες. Οι προσδοκίε επίσης και ότι ο τομέας αεροπορία θα κάνει περισσότερα από ότι απλώ και μόνο ε, την ανάπτυξη ε, ουδέτερος προς τον άνθρακα για το 2020. Και φυσικά δεν είναι μόνο το θέμα των εκπομπών, υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές ε, στις οποίες θα μπορούσε να επικεντρωθεί ο κλάδος για να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Για παράδειγμα, χρήση πλαστικών, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε από αυτού και πρέπει να πάμε και πέραν ε, της συζήτησης του Κορσία, να την προχωρήσουμε και άλλο και να είμαστε ε, πολύ πιο φιλόδεξοι. Και φυσικά υπάρχουν βιώσιμα καύσιμα αεροπορία και υπάρχουν κάποιοι που μας υποστηρίζουν και αυτό που έχει σημασία είναι να συνεχιστούν αυτές οι διαδικασίες αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε περισσότερα και θα πάμε πολύ παραπέρα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Α, ναι. Η ερώτηση του Αντιπροέδρου για τη γερμανική φορολόγηση και την αμερικανική επιστολή. Ε, φυσικά είναι βιομηχανία. Σίγουρα θα σταλούν τέτοιε επιστολέ και θα προσπαθήσουν να πιέσουν τα πράγματα και να πούμε ότι εμεί το ερμηνεύουμε έτσι. Εμεί όμω δεν το ερμηνεύουμε έτσι και θα το διευκρινίσουμε και σαφέστατα ότι αυτό δεν είναι ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εμεί τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που είπαμε και προηγουμένω ε, για τη σύμβαση του Σικάγο και το γεγονός ότι υπάρχει η ε, δυνατότητα λήψης αποφάσεων αυτόνομα πρέπει να το διευκρινίσουμε και στους διεθνείς μας εταίρους. Προφανώς και ο κλάδος θα συνεχίσει πάντα να αναζητά έναν τρόπο να πιέσει τα δικά του τα θέματα και φυσικά εμείς θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους εξηγήσουμε τι δεν μπορούν να κάνουν και τι μπορούν να κάνουν. Να πω λοιπόν ότι όπως είπατε θα απαντήσουμε και εμείς σε αυτό όταν τεθεί το ζήτημα σαφέστατα και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει καμία παραβίαση της ε, Συμφωνίας Μεταφορών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών που είναι και ένα από τα θέματα που έθιξαν εκεί. Και τώρα... Νομίζω ότι έγινε και μία παρατήρηση για τα εναλλακτικά καύσιμα και τις ε, ιδιότητες των ε, ε, αεροπορικών μεταφορών, ε, να σας πω ότι ένα σχέδιο offsetting, ε, τα ρώτησε ο κύριος Γουάλαγκ αυτά, είναι οικονομικά βιώσιμο μόνο σε τομείς στους οποίους είναι πολύ εύκολο να έχουμε μειώσει σε τεχνικό επίπεδο και επομένως να μειώσουμε και το κόστος. Αλλά η αποτελεσματικότητα ενό τέτοιου προγράμματος εξαρτάται και από την ποιότητα του προγράμματος ε, που χρηματοδοτείται για να μειωθούν οι εκπομπές. Και φυσικά υπάρχει και τεχνικό συμβούλιο στον ΑΙΚΟ, στο οποίο έχουμε ανεξάρτητους υψηλού επίπεδου εμπειρογνώμονες που εξετάζουν τέτοια προγράμματα τα οποία ε, θα αναγνωριστούν τον Ιούλιο από το Κορσία και όλα αυτά θα πρέπει να ξεκινήσουν από τα προγράμματα τα οποία αναγνωρίστηκαν από το Κορσία. Υπάρχουν ε, εκθέσεις προόδου οι οποίες προβλέπονται καθώς και αξιολογήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να υπάρχει και η απαραίτητη ποιότητα. Όσον αφορά λοιπόν την ε, πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου, θα τη λάβει υπόψη το Συμβούλιο του ΑΙΚΑΟ για να λάβει υπόψη ε, βάση των ε, κριτηρίων επιλεξιμότητων των μονάδων εκπομπών που έχουν επιλέξει εμπειρογνώματος και αυτό θα μας εξασφαλίσει ότι οι εκπομπές θα αντισταθμίζονται με προγράμματα επιτόπου που θα καθορίζουν μόνιμες και πολύ συγκεκριμένε επαληθευμένες μειώσεις αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου ε, για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και τις υποχρεώσεις μετριασμού. Όλα αυτά θα είναι σχετικά αυστηρά. Εμείς συμμετέχουμε σε συζητήσεις, οι εμπειρογνώμονες μας συμμετέχουν σε συζητήσεις και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, έχουμε παρουσία εκεί και να συνεχιστεί αυτό. Ένα τελευταίο σημείο, κριτήρια βιωσιμότητας για βιώσιμα καύσιμα ε, για τις αεροπορίες. Για το πιλωτικό στάδιο 2021-2023 έχουν εγκριθεί τρία κριτήρια που εγγυώνται ελάχιστον 10% εξοικονόμηση εκπομπών και ε, τα βιοκαύσιμα ε, προέλευσης από ζωοτροφές δεν θα είναι ε, υψηλής χρήσης άνθρακα. Ε, ζητήθηκε να εγκριθούν 12 κριτήρια βιωσιμότητα στον ΑΙΚΑΟ, τα υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συζητηθούν στον επόμενου μήνε και φυσικά είναι εγγύηση ότι δεν ε, θα κάνουμε κάτι με τη βιώσιμη αεροπορία, κάτι το οποίο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο. Ευχαριστώ που μακρηγόρησα, το ξέρω, αλλά μου ζητήσατε να είμαι συγκεκριμένο. Για το δεύτερο γύρο τώρα έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Ε, Αντέλη, λοιπόν καταρχήν και μετά Μαρτινόσικ και μετά θα ακούσουμε απαντήσεις. Ευχαριστώ ε, κύριε Γενική Διευθυντά. Είπατε μόλις τώρα ότι θέλετε να κάνουμε περισσότερα και να πάμε πιο μακριά. Είναι θετικό το το ακόμα αυτό, αλλά εμείς είμαστε εκνευρισμένοι γιατί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην, στον επίγοντα χαρακτήρα αυτής της ανάγκης του να μειωθούν δηλαδή οι εκπομπές ε, από όλου του τομείς αφενός και με την συμπεριφορά από την πλευρά των επιχειρήσεων αφετέρου. Δηλαδή βλέπουμε οι επιχειρήσεις να ακολουθούν μια τακτική τύπου όλα έχουν όπως είχαν, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουν γίνει ε, τα κατάλληλα βήματα ώστε να ελεγχθούν οι εκπομπές αυτές από την πλευρά των επιχειρήσεων. Εγώ έχω έρθει σε επαφή με επιχειρήσει και μου λένε ότι συχνά ε, είναι ο αποδιοπομπαίο τράγο. Αλλά δεν ε, θεωρώ πω συμβαίνει αυτό, γιατί εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε σοβαροί ω προ το στόχο που έχουμε θέσει να έχουμε μηδενικέ εκπομπέ ανθρακά στο 2050. Το γεγονό ότι λοιπόν ο ΤΟΙΚΑΟ προσπαθούσε να μπλοκάρει περιοχέ και χώρε που θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω είναι κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Θα ήθελα επίση να είχα δει μια πιο κατηγορηματική, πιο ισχυρή στάση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή τη Ένωσης και για τη δική μου άποψη θα πρέπει να εκφράσει όχι μόνο προφορικέ αντιρρήσει, αλλά να προβεί σε πραγματική αντίρρηση, δηλαδή γραπτή η οποία μπορεί, μπορεί να αποτελέσει και ένα σημείο αναφορά στο μέλλον, σε ό,τι αφορά δηλαδή τι δυνατότητε ε, που θα μπορεί να έχει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώνει τι εκπομπέ τη μέσω του ETS. Και αναφερθήκατε εσεί ειδικότερα στο ζήτημα του offset, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε τι εκπομπέ του χώρου τη αεροπορία. Εκπομπέ οι οποίε έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και αν το κάνουμε αυτό, δηλαδή έχουμε ένα τέτοιο σύστημα offset, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο των μηδενικών εκπομπών του 2050. Άρα λοιπόν θα ήθελα να σα παρακαλέσω να είμαστε ξεκάθαροι ω προ το στόχο του ότι δεν μπορούμε, δεν είναι πανάτια το να δεν μπορεί να λύσει το όλο πρόβλημα το να έχουμε carbon offsetting, θα πρέπει να ε, λάβουμε περαιτέρω μέτρα. Ο κύριο Ευχαριστώ. Ναι, είναι σαν να ακούμε λόγια από έναν άλλο παράλληλο κόσμο. Δηλαδή, έως το 2030 πρέπει να έχουμε μειώσει κατά 55% ε, τα αέρια του θερμοκηπίου αλλά ε, έχουν αυξηθεί κατά παραπάνω από 25% τα τελευταία χρόνια εκπομπέ τη αεροπορία. Οπότε είναι κάτι το εντελώ αντίθετο. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, το επίπεδο δέσμευση για το Κόρσια και το πόσο φιλόδοξοι θέλουμε να είμαστε, νομίζω πω πρέπει να είναι αντίστροφη η πορεία. Δηλαδή, θα πρέπει καταρχήν να υπάρξει μια δέσμευση φιλόδοξη σε ό,τι αφορά του στόχου και μετά το Κόρσια θα πρέπει να κληθεί να ε, βοηθήσει στην ε, επίτευξή του. Δηλαδή, αν ο πλανήτη είναι νεκρός, τότε κανένα δεν μπορεί να έχει αναπτύσσει και δεν, σε τίποτα δεν ωφελεί η αεροπορία και νομίζω αυτό μερικέ φορέ το ξεχνούν και επιχειρήσει το ξεχνά και η Επιτροπή. Δηλαδή, ακούμε τώρα εδώ ότι ο ΕΚΑΟ ξεκινάει τώρα τι συζητήσει ω προ το πότε ε, φτάσουμε κάποια στιγμή σε κάποιους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών. Μα δεν είμαστε το 1999, το 2019 είμαστε. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα πότε σκοπεύετε να υπάρξουν συγκεκριμένοι στόχοι και σε επίπεδο ΙΚΑΟ αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του συστήματο εκπορία εκπομπών του ΟΕΤΕ. Και δηλαδή, ποιοι θα είναι οι στόχοι για το ETS ε, σε ό,τι αφορά την αεροπορία αντί να δίνουμε ελεύθερες πιστώσεις. Δηλαδή, πότε θα υποχρεώσουμε τις αεροπορικές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται επί ίσης όλες με όλους τους υπολείπους. I can save. Ε, κυρία Πάουλος λέω ότι καλύφθηκα ήδη εγώ από τον κύριο Χόζεκ, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι από την πλευρά μου. Πρόεδρος, δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, οπότε έχετε το λόγο, κύριε Γενική Διευθυντά, για δύο-τρία λεπτά ακόμα που μας απομένουν για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτές τις ερωτήσεις και για αυτά τα σχόλια και για το γεγονός ότι εδώ τα μέλη του Κοινοβουλίου θέλουν να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Τα όσα ανέφερε η κυρία Ντάλη, νομίζω πως καταρχήν μας βρίσκουν ε, σύμφωνο στο ότι δηλαδή δεν μπορεί να ακολουθήσει ε, ο επιχειρηματικός κλάδος την ίδια τακτική, την ίδια πρακτικές με αυτές που εφήρμοζε μέχρι τώρα. Νομίζω πως αυτό είναι ξεκάθαρο για όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορίας. Αλλά κατά τη δική μου άποψη, ε, χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να συνειδητοποιήσει και ο αεροπορικό τομέα ότι πράγματι δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί ο τρόπο λειτουργία αυτού του κλάδου έτσι όπω ε, ήταν μέχρι τώρα. Δηλαδή έχει αρχίσει ο κλάδο να το παίρνει πολύ πιο σοβαρά αυτό το ζήτημα υπόψη του. Τώρα σε ό,τι αφορά το, τον ΕΚΑΒ. Πρόκειται για ένα σώμα των Ηνωμένων Εθνών, για έναν οργανισμό ε, στον οποίο συμμετέχουν 193 διαφορετικές χώρες και κατά συνέπεια η πρόοδος η οποία επιτυγχάνεται δεν γίνεται με αλματώδεις ρυθμούς, γίνεται σταδιακά αργά και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ε, πιέζουμε έτσι ώστε να γίνονται κάποια βήματα έστω και μικρά. Και γι' αυτό ακριβώς πιέζουμε ως προς το να ε, είναι πράγματι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα ένας βασικός στόχος και ο νέος πρόεδρος της ΕΚΑΟ θα πρέπει να τονίσω ότι πράγματι το έχει θέσει ως προτεραιότητα αυτό το ζήτημα και έχει ε, αυξηθεί ακριβώς η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε σύγκριση δηλαδή με το πώς είχαν τα πράγματα πριν από κάποια χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το carbon offsetting, ε, προφανώς δεν επαρκεί αυτό για να φτάσουμε τελικά στι μηδενικέ εκπομπέ. Δηλαδή θα χρειαστεί κάποια στιγμή να έχουμε πραγματική μείωση των εκπομπών στον αεροπορικό τομέα και θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιε ε, λύσει θα βρεθούν στο πλαίσιο του Green Deal. Ε, και ακριβώς αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ιδέα που αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά τα βιώσιμα καύσιμα ε, για την αεροπορία. Εάν δηλαδή μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τέτοιου είδου καύσιμα μπορούν να αποτελέσουν ένα πραγματικό υποκατάστατο, πλήρε υποκατάστατο τη κυροζήνη μέσω και μακροπρόθεσμα, τότε θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε περαιτέρω στο στόχο των μηδενικών εκπομπών. Τώρα, σε ό,τι αφορά και πάλι το Κόρσια, να πω κάτι ακόμα. Τελευταίο σχόλιο από την πλευρά μου, Πρόεδρε. Είναι λοιπόν το εξή, ότι σύμφωνα με τον υπολογισμό που έχει γίνει, Ε, θα μπορούσαμε να έχουμε μείωση, αν εφαρμοστεί σωστά το κόρσια, ε, κατά 3,5 δις ε, τόνους διοξιδίου του άνθρακα σε επίπεδο εκπομπών δηλαδή και θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν και 40 δις έως το 2035. Άρα λοιπόν το Κόρσια μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει ουσιαστικά στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο, θα έχουμε τη δυνατότητα στο πλαίσιο τη ανακοίνωση για τον Green Deal από την πλευρά τη Επιτροπή να ξανασυζητήσουμε αυτό το ζήτημα, αφού στο πλαίσιο εκείνη τη ανακοίνωση ο αεροπορικό τομέα θα είναι εκείνο που θα μα απασχολήσει περισσότερο. Είτε το, δηλαδή τον ε, εξετάσουμε από φορολογική άποψη, ε, είτε τον εξετάσουμε από την πλευρά του συστήματο εμπορίου εκπομπών, είτε και από άλλε οπτικέ γωνίε. Σα ευχαριστώ λοιπόν και πάλι κύριε Γενική Διευθυντά το γεγονό ότι είχαμε μια πολύ ανοιχτή και διαφανή συζήτηση εδώ με εσά, με την Γενική Διευθύνση μου και βέβαια σε μερικέ. Ε, μέσα στι επόμενε μέρε θα έχουμε μια νέα ακρόαση του Πετρόπου Μεταφορών. Έτσι και πάλι λοιπόν θα έχουμε εκεί τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ τη Επιτροπή για τα σκληρά ερωτήματα που μου έθεσαν και τα επικριτικά του σχόλια αλλά πραγματικά ε, χαίρομαι πάντοτε που συζητώ εδώ μαζί σε αυτά τα ζητήματα έτσι ώστε να προωθήσουμε περαιτέρω αυτά τα θέματα και θα είμαι και μελλοντικά πάντοτε στη διάθεσή σας. Uh, Ωραία, συνεχίζουμε και περνάμε στο δεύτερο τμήμα της σημερινής μας συνεδρίασης. Καλωσορίζω εδώ λοιπόν τους επικεφαλείς των οργανισμών ε, που έχουν ε, θέματα, που είναι αρμοδιότητα, έχουν καθήκοντα που είναι αρμοδιότητες της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Λοιπόν, Θα οργανωθούμε ως εξή. Θα αρχίσουμε με μία δεκάλεπτη εισαγωγή του κυρίου Αντρέα Άμον, που είναι ο πρόεδρος του ECDC, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, και μετά θα ακούσουμε την ΕΚΑ, την ΕΜΑ, την ΕΦΣΑ και την EA Έχουμε τα θέματα υγείας, τα θέματα του περιβάλλοντος και τα δύο συνδέονται βέβαια πολλές φορές και μετά φυσικά θα ε, μπορούμε να έχουμε ερωτήσεις πρώτα απ' όλα από αυτούς που είναι τα σημεία επαφής. Αρχίζουμε λοιπόν με τη δεκάλεπτη παρουσίαση για το συνολικό σύστημα των οργανισμών αυτών. Από, τον κύριο, από την κυρία Μον, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τους τέσσερις οργανισμούς μας. Είναι η δεύτερη φορά μάλιστα που είμαστε εδώ και έχουμε αυτή την ευκαιρία στην αρχή της θητείας ε, της Επιτροπής ΕΝΒΗ να σας συστηθούμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Πρόεδρο και την Γραμματεία που βοήθησαν σε αυτό. Είμαι λοιπόν η Διευθύντρια του ECDC, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Τώρα όμως σας μιλάω ως Πρόεδρος και των πέντε ε, οργανισμών που αποτελούν ένα δίκτυο γιατί και οι πέντε εξετάζουν ε, θέματα που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Εμείς ε, φροντίζουμε να βοηθήσουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών με τη δικιά μας πραγματογνωμοσύνη, είτε τεχνική είτε επιστημονική. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω λιγάκι εδώ τι κάνουν για τους πολίτες οι οργανισμοί αυτοί για να μην τα ξαναπούμε κάθε φορά με τις παρουσιάσεις των επιμέρους οργανισμών. Στόχος μας λοιπόν είναι να χρησιμοποιηθεί η συνδυασμένη πραγματογνωμοσύνη μας και η γνώση μας η τεχνική και η επιστημονική που είναι διαθέσιμη για σας τους ευρωβουλευτές. Η πραγματογνωμοσύνη μας μπορεί να βοηθήσει να υλοποιηθούν οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως είναι για παράδειγμα η βιώσιμη στόχη ανάπτυξης, η στόχη του 2030 δηλαδή, μηδενική ρήπανση και Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Και ο πρόεδρος, ο κύριος Καλφέν, το είπε όταν έγινε πρόεδρος Επιτροπής αυτής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη φιλοδοξία σε όλους τους τομείς που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ΕΝΒΗ και εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας για τη φιλοδοξία αυτή. Τώρα και οι πέντε οργανισμοί ε, δουλεύουν για θέματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πρόκειται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, προστασία του περιβάλλοντος, να καταστεί περισσότερο ασφαλής η Ευρωπαϊκή Ένωση με περισσότερη υγεία και περισσότερο ανταγωνιστική. Και εδώ σε μία εικόνα έχουμε βάλει το τι αντιπροσωπούμε και το ε, τι κάνουμε. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει αυτό το σύννεφο λέξεων. Εδώ θα δείτε διάφορες λέξεις κλειδί, όπως είναι η επιστήμη, η υγεία, η ασφάλεια, η ευρωπαϊκή πραγματογνωμοσύνη, αλλά και κάποιες άλλες λέξεις που έχουν να κάνουν περισσότερο με, με τον έναν ή τον άλλον οργανισμό, όπως είναι τα φάρμακα, τα χημικά, το περιβάλλον, τα τρόφιμα και οι ασθένειες. Τώρα, οι οργανισμοί μας λειτουργούν βέβαια διαφορετικά, αλλά έχουν και κοινά σημεία στη λειτουργία τους. Όλοι ε, λειτουργούμε με ανεξαρτησία και με διαφάνεια και συμμετέχουν ε, στο έργο μας και τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι η κοινωνία των πολιτών, με κυβερνητικέ οργανώσεις, καταναλωτές, ασθενείς, αγρότες ε, και γενικότερα το κοινό. Εμείς θέλουμε να προσφέρουμε στοιχεία επιστημονικά, γνωμοδοτήσεις που βασίζονται σε στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του κοινού στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Επίσης, ε, δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε και με τις αρχές και με εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις προκειμένου το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βασίζεται σε επισημονικά δεδομένα. Τώρα γνωρίζουμε ότι εσείς έχετε πολλές και διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες, την βιοποικιλότητα, την κυκλική οικονομία, τη δημόσια υγεία, την ασφαλεία τροφίμων, η ποιότητα του αέρα και των υδάτων, ε, προστασία από τα χημικά, τα φυτοφάρμακα κλπ. Εμείς λοιπόν Χρησιμοποιούμε την καλύτερη επιστημονική γνώση από τις χώρες μέλη και την πραγματογνωμοσύνη και διασφαλίζουμε ότι οι γνωμοδοτήσεις μας βασίζονται στα καλύτερα δεδομένα. Και οι γνωμοδοτήσεις μας βοηθούν εσάς να πάρετε αποφάσεις και μπορούμε έτσι να σας προσφέρουμε εμείς μια ευρία ευρωπαϊκή προπτική. Τώρα, όσον αφορά τι σωστέ πολιτικέ αποφάσει, χρειάζεται βέβαια και αποτελεσματικότητα. Δεν υπάρχει ούτε χρόνο για χάσιμο, ούτε χρήμα. Έτσι λοιπόν, εφόσον δουλεύουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εσεί που λαμβάνετε τι αποφάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, γίνονται περισσότερο αποτελεσματικοί. Για πολλού από εμά, οι χώρε ε, μέλη ε, συμμετέχουν και στα διοικητικά μας ε, συμβούλια και επίσης έχουμε και ευρωβουλευτές και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εδώ σήμερα. Οι προτερότητες μας έχουν ως στόχο να κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών μας. Συνεισφέρουμε λοιπόν σε αυτό το στόχο όλοι οι οργανισμοί αυτοί και επίσης μπορούν να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας οι καταναλωτές γιατί εμείς διασφαλίζουμε κοινέ προδιαγραφές για αυτούς. Οπότε, οι οργανισμοί αυτοί είναι εδώ για να σας στηρίξουν. Και το κάνουν με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Για παράδειγμα, την τεχνική μας και επιστημονική μας γνώση τη μοιραζόμαστε ε, μαζί σας για την προετοιμασία της πολιτικής που εκπονείτε. Σας παρουσιάζουμε τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και επίσης κατά την υλοποίηση της νομοθεσίας επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί στηρίζουμε τις χώρες μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές υπό το πνεύμα του νομοθέτη. Επίσης, κατά την αξιολόγηση των πολιτικών σας και των προγραμμάτων σας, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε δίνοντας συγκεκριμένα και πρακτικά παραδείγματα, δίνοντας feedback με τα στοιχεία τα οποία εμείς συλλέγουμε. Επίσης, βοηθάμε για να απαντηθούν οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και βοηθάμε και για την εκπόνηση ψηφισμάτων εφόσον εσείς μας δείστε ή εκθέσεων εφόσον μας το ζητήσετε. Συνεπώς, επίσης λογοδοτούμε σε εσά. Υπάρχει διαδικασία απαλλαγή και υπάρχουν και οι αιτήσιε ακροασει των διευθυντών των οργανισμών αυτών. Εμείς, όπως βλέπετε και σε αυτή τη διαφάνεια, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες και τις προτεραιότητές σας. Και έτσι όλοι μας προσπαθούμε να προχωρήσουμε για αυτά τα θέματα, να τα αναλύσουμε παρετέρω και να σας δώσουμε παραδείγματα και τις συνεργασίες μας. Σίγουρα έχετε πάρει μέχρι τώρα τις πληροφορίες για το πώς λειτουργούμε, αλλά έχουμε ετοιμάσει και ψηφιακά κάποιες πληροφορίες γιατί δεν θέλουμε να τυπώνουμε χαρτί. Οπότε θα τα βρείτε στις ιστοσελίδες μας σε ψηφιακή μορφή. Τέλος εδώ είναι οι διευθύνσει μας που υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής ΕΝΒΗ και είμαστε στη διάθεσή σας. Μην διστάζετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για να μας ζητήσετε συνεργασία. Ε, θέλουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας και όχι μόνο μέσω των ευρωβουλευτών που αποτελούν τα σημεία επαφή μα. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ όλου και επαναλαμβάνω αυτό που είπε και ο πρόεδρο, ότι οι πέντε οργανισμοί προσφέρουν στο τέλο τη συνεδρίασης αυτή ένα μικρό ποτό και σα το όλοι Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα περάσουμε στις παρουσιάσεις λοιπόν λοιπόν την ΕΚΑ, την ΕΦΣΑ και την ΕΕ πρώτα απ' όλα. Παρακαλώ, εσείς, η ΕΚΑ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων. Yes, thank you very much. Um, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, μέλη. Θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός χημικών προϊόντων συνεργάζεται σε μεγάλο βαθμό με τους εταίρους, δηλαδή τα κράτη-μέλη, την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, αλλά και τους ε, διάφορους ε, αρμόδιους ε, φορείς, τους stakeholders, δηλαδή που εκπροσωπούν από την πλευρά τους τις επιχειρήσεις, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ειδικότερα τις περιβαλλοντικές, αλλά και άλλες, όπως για παράδειγμα εκείνες της προστασίας των ζώων. Και βέβαια ο βασικός στόχος είναι η ασφαλής χρήση των χημικών προϊόντων. Πώς το επιτυγχάνουμε αυτό μέσω της εφαρμογής διαφορετικών νομικών πράξεων, νομοθεσίας δηλαδή ε, ευρέω σπάσματο σε ό,τι αφορά την ασφαλή αυτή χρήση. Τα βλέπετε εδώ στη διαφάνεια, δεν θα αναφερθώ λεπτομέρω. Αλλά ο στόχο είναι η ασφάλεια. ασφάλεια δηλαδή των εργαζομένων, των καταναλωτών όταν χρησιμοποιούν τα ενόγω χημικά προϊόντα, αλλά και των πολιτών οι οποίοι χωρίς να το επιθυμούν, αν επιθυμούνται δηλαδή, εκτίθενται σε αυτά τα χημικά προϊόντα, αλλά και το περιβάλλον το οποίο εκτίθεται σε αυτά. Έτσι λοιπόν, με το δικό μας τρόπο συνεισφέρουμε στους τομείς πολιτικής της ε, βιοποικιλότητας, της προστασίας των υδάτων, ε, της ε, ατμόσφαιρας, δηλαδή της ποιότητας του αέρα και παρότι προσανατολιζόμαστε ειδικότερα σε εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε και κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν την παγκόσμια ατζέντα σε ό,τι αφορά τα χημικά προϊόντα. Επίση, μέσω τη δουλειά που κάνουμε ε, προ όφελο τη ασφάλεια, συνεισφέρουμε σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά τη Ένωση, καθώ εξασφαλίζουμε αυτόν τον τρόπο ένα θεμητό και δίκαιο ανταγωνισμό. Έτσι, με αυτήν την ασφάλεια δηλαδή την οποία εξασφαλίζουμε στην εσωτερική αγορά, επιτρέπουμε ε, στην ε, στον κλάδο των καινοτόμων φαρμάκων να, και χημικών να ανθεί και με αυτόν τον τρόπο βέβαια προωθούμε τις ε, καινοτομίες γενικότερα στον βιομηχανικό ε, τομέα και τον χώρο της μεταποίησης. Και μέσω ακριβώς αυτής της ε, εξασφάλισης της ασφάλειας συμβάλλουμε στην ανταγωνιστικότητα όχι μόνο αυτών των επιχειρήσεων, δηλαδή του συγκεκριμένου κλάδου των χημικών προϊόντων, αλλά και γενικότερα των επιχειρήσεων της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της ε, προστασίας της ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας, ε, της καινοτομίας ε, στον εσωτερικό, στην εσωτερική αγορά, έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία, το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο μας επιτρέπει συνέργειες ανάμεσα στις διαφορετικές νομοθεσίες. Έτσι έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα και ταχύτερη εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας. Και αυτό πάλι βέβαια με τη σειρά του προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την εύρυθμη λειτουργία στην εσωτερική αγορά. Ταυτόχρονα όμω με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την περισσότερη αρμονική αν θέλετε συνύπαρξη, την συνέργεια αλλά και την συνέπεια ανάμεσα στις διαφορετικές διατάξεις ε, τη διαφορετική νομοθεσία στου διαφορετικού διαφορετικούς Βέβαια όλη μας η εργασία βασίζεται στο προσωπικό μας, ε, στην ε, εμπειρία μας. Αλλά εδώ ειδικότερα για να αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας βασιζόμαστε στη μεγαλύτερη βάση δεδομένων παγκοσμίω σε ό,τι αφορά τα χημικά προϊόντα. Και χρησιμοποιείται όχι από εμάς, αλλά και από όλους στην Ένωση οι οποίοι εργάζονται ή παράγουν χημικά προϊόντα. Δηλαδή και εδώ οι επιχειρήσεις ε, έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων και με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζονται σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητά τους αλλά και την κοινοτομία τους. έχουμε από εκεί και μετά πολύ συγκεκριμένε αρμοδιότητε εδώ, δηλαδή διαχείριση των δεδομένων, αξιολόγηση των χημικών προϊόντων, διαχείριση των κινδύνων των χημικών προϊόντων και αξιολόγηση των κοινών οικονομικών επιπτώσεων τη χρήση αλλά και τη διαχείριση των λόγω χημικών προϊόντων. Οι εν λόγω λοιπόν αρμοδιότητε είναι αρμοδιότητε τι οποίε αναλαμβάνουμε, γνωρίζοντα πολύ καλά ότι οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν σε σχέση με αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή και το Ευρωβαρόμετρο και οι εθνικέ οικομετρήσει το έχουν καταδείξει αυτό επανειλημμένα και έτσι λοιπόν προσπαθούμε ένεργα να διασκεδάζουμε αυτέ τι ανησυχίε των πολιτών μα μέσω τη ανάληψη αυτών των καθηκόντων από τη δική μα πλευρά, αλλά και αυξάνοντα την ευρύτερη γνώση για τα χημικά προϊόντα, αλλά και την πιο εξειδικευμένη χρήση του Αλλά Βέβαια, προωθούμε ταυτόχρονα την ασφαλή του χρήση και αυξάνουμε τη διαφάνεια έτσι ώστε οι πολίτε μα να γνωρίζουν ότι ό,τι πράττουμε από δική μας πλευρά, δηλαδή σε επίπεδο αυτή τη διαχείριση ε, των χημικών προϊόντων, γίνεται με βάση αξιόπιστες επιστημονικέ πληροφορίε. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθούμε εμεί να κάνουμε είναι να είμαστε υπηρεσία η οποία αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι ε, της διαχείρισης των χημικών προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να συμβάλλουμε στο να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση όταν εσείς αποφασίσετε ότι θα πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι για να αναλάβουμε δράση όταν θα χρειαστεί αυτό να το κάνουμε από τη δική μας πλευρά, όταν θα μας το ζητήσετε. Και με στις επόμενες δύο διαφάνειες θα σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Προφανώς λοιπόν υπάρχει αυτή η ατζέντα για την κυκλική οικονομία, ε, η οποία θεωρούμε πως ε, θα προωθηθεί ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τρέχουσας ε, θητείας Κοινοβουλίου και τη επιτροπή ε, και υπάρχει και το ζήτημα του Green Deal που θα αποτελέσει δηλαδή μια ευρύτερη γενικότερη προτεραιότητα όπως έχει ήδη αναφερθεί από την ε, νέα Επίτροπο, ε, πρόεδρο της Επιτροπής. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε εμείς ό,τι αφορά ειδικότερα την κυκλική οικονομία, κατά κύριο έχουμε να κάνουμε κυρίως με την επαναχρησιμοποίηση, δηλαδή την κυκλική χρήση των προϊόντων. Αλλά όλα τα προϊόντα ε, βασίζονται ή συναποτελούνται από χημικά. Άρα λοιπόν ό,τι συμβαίνει σε αυτό το τομέα πάντοτε εμπλέκει και τον έκα γιατί ουσιαστικά όταν κάνουμε λόγο για προϊόντα κάνουμε λόγο για χημικά προϊόντα. Αλλά και η καινοτομία από τον κλάδο χημικών προϊόντων μας θα αποτελέσει κινητήριο ε, δύναμη για την αντιμετώπιση μιας σειράς κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή με τεχνικές λύσεις μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής. Αλλά η εν λόγω λύσεις βέβαια θα πρέπει να είναι ασφαλείς και εδώ ακριβώς ερχόμαστε να παίξουμε το δικό μας ρόλο ως οργανισμός χημικών προϊόντων. Εδώ λοιπόν συμβάλλουμε με τις ε, γνώσεις μας, με τις με την ικανότητα που έχουμε, ακριβώς για να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία και να συμβάλλουμε στην θέσπιση, στη διαμόρφωση ενός Green Deal. Και για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε οργανώσει με τέτοιο τρόπο την, ε, ε, τον οργανισμό μας, ο οποίος θα μας επιτρέψει να αναλάβουμε πολύ ευκολότερα νέα καθήκοντα και να τα εντάξουμε ε, στη δουλειά που κάνουμε αυτή την περίοδο σε σχέση με άλλα είδη νομοθεσία. Έτσι ώστε δηλαδή να είμαστε ταχύτεροι σε ό,τι αφορά την ένταξη αυτών των νέων καθηκόντων στι ευρύτερε εργασίε μα και διασφάλιση τη συνέπεια. Και επίση ταυτόχρονα εξετάζουμε από θεμική άποψη ε, τη δυνατότητα του να αξιολογούμε, ε, να εξετάζουμε δηλαδή όχι συγκεκριμένες ουσίες, συγκεκριμένα χημικά προϊόντα, αλλά ομάδες ουσιών. Και μέχρι τα τέλη του επόμενου χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει αυτή την πρώτη διαδικασία. Εδώ, σε αυτή την διαφάνεια τώρα βλέπετε το προσωπικό μας εδώ, γύρω στο 1 τρίτο εμφανίζεται σε αυτή τη φωτογραφία και βέβαια η εμπειρία όλων αυτών των ε, συνεργατών μας είναι εκείνη στην οποία βασιζόμαστε σε ό,τι αφορά την βιώσιμη χρήση ε, των χημικών προϊόντων προ όφελο και των πολιτών μα, αλλά και του περιβάλλοντος. Αυτά λοιπόν από τη δική μου πλευρά σε πλαίσιο αυτών των πέντε παρουσιάσεων που θα ακούσετε από, ε, από τους πέντε διαφορετικούς οργανισμούς. Ευχαριστώ. Θα πάμε τώρα στην ΕΦΣΑ. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Με ιδιαίτερη χαρά θα σας παρουσιάσω τώρα την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων. Είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην Ιταλία, στην Πάρμα, με 500 ανθρώπους προσωπικό. Και βλέπετε τι κάνουμε εδώ κάτω αριστερά στην διαφάνεια αυτή. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε την επιστήμη για ασφαλή τρόφιμα. Βασιζόμαστε στην επιστήμη για ασφαλή τρόφιμα. Αυτό κάνουμε. Λέμε ότι αν δεν είναι ασφαλές, δεν είναι τρόφιμο. Οπότε όλα ξεκινούν με την ασφάλεια τροφίμων. Αλλά την ασφάλεια τροφίμων βέβαια τη βάζουμε σαν γενικότερο πλαίσιο διατροφής, υγείας και βιωσιμότητας. Οπότε ασφαλή τρόφιμα είναι το σημείο κίνησης, αλλά πρέπει να το δούμε στο γενικότερο πλαίσιο της υγείας και της βιωσιμότητας. Πόσο μπορεί δηλαδή το τρόφιμο αυτό να παραχθεί και στο μέλλον θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα ε, τρόφιμα για 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Πώς θα το κάνουμε αυτό με βιώσιμο τρόπο και προστατεύοντας την υγεία. Χρειαζόμαστε την επιστήμη, γι' αυτό λέμε εμπιστευόμαστε την επιστήμη για την ασφάλεια τροφίμων. Είμαστε δηλαδή επιστημονικοί σύμβουλοι των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Είμαστε σύμβουλοι σας ουσιαστικά για να βοηθήσουμε οι πολιτικές αποφάσεις να ληφθούν βάση δεδομένων και επιστημονικών στοιχείων. Πρόσφατα στο Ευρωβαρόμετρο υπήρχε ερώτηση τι σκέφτεστε όταν πηγαίνετε να ψωνίσετε, ποια είναι η κυριότερη ανησυχία σα. Και η ασφάλεια τροφίμων δεν ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία των Ευρωπαίων καταναλωτών, ήταν ε, μία από τι πρώτε 5. 22% των ανθρώπων θεωρούν ω κύρια ανησυχία του στην ασφάλεια τροφίμων όταν πηγαίνουν να ψωνίσουν. Κάτι το οποίο είναι θετικό γιατί δείχνει ότι το σύστημα, οι χώρε μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κλάδο των τροφίμων αλλά και εμεί κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Λοιπόν, τι κάνουμε. Εδώ το βλέπετε. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά κάνουμε πράγματα για πολλά και διαφορετικά νομοθετήματα. Ε, προσφέρουμε δηλαδή την επιστημονική γνώση για τους διαχειριστές και για αυτούς που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις για την ασφάλεια τροφίμων και την κάνουμε με την ιδέα από το χώμα στο στόμα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι δηλαδή μια προσέγγιση που πιστεύω ότι πρέπει να τη δείτε ακριβώς στο γενικότερο πλαίσιο της ασφαλείας ε, τροφίμων και των τροφίμων, γιατί πρόκειται για ένα βιολογικό σύστημα, ένα κοινωνικό σύστημα και ένα οικονομικό σύστημα ε, που θα πρέπει να τροποποιηθεί τα επόμενα χρόνια για να έχουμε ασφαλή, υγιή και βιώσιμα τρόφιμα. Επίσης έχουμε και τον ιδρυτικό μας κανονισμό που μας ζητάει να επικοινωνούμε ε, τους κινδύνους. Η δέσμευσή μας αυτή δηλαδή είναι μια νομική μας υποχρέωση και είναι καλή, είναι θετικό που υπάρχει, ώστε με ανεξαρτησία έγκαιρα να ενημερώνουμε για τους κινδύνους την διατροφική αλυσίδα. Να ενημερώνονται και οι καταναλωτές αλλά και οι διαχειριστές και τα μέσα ενημέρωσης. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε επίση επιστημονική συνεργασία. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αν δεν έχουμε συνεργασία με τι χώρε μέλη. Οι χώρε μέλη είναι που μα δίνουν του εμπειρογνώμονέ του. Είναι αυτοί που είναι στα πάνελ μα και χωρί αυτή την ευρωπαϊκή συνεργασία δεν θα μπορούσε η ΕΦΣΑ να κάνει τη δουλειά τη. Εδώ. Σε τι βάση εργαζόμαστε, τι μας δίνει την ενέργεια να δουλεύουμε σε καθημερινή βάση για μεγαλύτερη ασφάλεια στα τρόφιμα. Είναι επιστημονική αριστεία πρώτα απ' όλα. Έχουμε την υποχρέωση αλλά και τη φιλοδοξία να σας προσφέρουμε την ε, καλύτερη επιστημονική γνώση και συμβουλή. Μιλάμε για την καινοτομία επίσης στην ε, αξιολόγηση κινδύνου γιατί η καινοτομία είναι συνεχής στον κλάδο των τροφίμων και εμείς πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα λάβουμε υπόψη μας τα νάνο υλικά, ε, τους ε, ορμονικούς διαταράχτες κλπ. κλπ. Χρειαζόμαστε λοιπόν την συνεργασία αυτή, είναι στο DNA του οργανισμού μας. Και οι τελευταίες μας αρχές είναι η ανεξαρτησία, γιατί έχουμε και εδώ νομική υποχρέωση να προσφέρουμε ανεξάρτητη επιστημονική ε, γνώμη. Η επιστήμη είναι αυτή που σας επιτρέπει να πάρετε τις σωστές αποφάσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιωσιμότητα. Και όλα αυτά τα κάνουμε με έναν ανοιχτό τρόπο. Είμαστε ανοιχτοί και τι σημαίνει αυτό. Έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, τη διαφάνεια και δεύτερον τη δέσμευσή μας. Και είμαστε ευγνώμονες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με τη νέα ρύθμιση για τη διαφάνεια που εγκρίθηκε πριν από μερικούς μήνες η ΕΦΣΑ αναλαμβάνει νέα καθήκοντα αλλά και νέες ε, πηγές, νέους σπόρους. Και γι' αυτό σας ζητάμε να μας βοηθήσετε στις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο οι πόροι που προβλέπονται να ελοπιθούν, Γιατί αυτοί είναι οι πόροι και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνουν θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε με έναν τρόπο με περισσότερη διαφάνεια και συμμετοχή όλων στις επιστημονικές μας αποφάσεις. Τέλος, για ποιον δουλεύουμε. Έχουμε τέσσερις πελάτες, να το πω έτσι. Το μεγαλύτερο έργο μας ε, μας το ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την ΕΦΣΑ. Μάλιστα αυτή την εποχή δουλεύουμε ε, για πράγματα που οποία μας έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ένα είναι η υγεία των μελισσών. Κοιτάμε διάφορου παράγοντες που επηρεάζουν ε, του επικονιαστές όπως επίσης κάτι και για τα κουνέλια. Έχει να κάνει με την προστασία των ζώων. Θέλουμε να προσφέρουμε επιστημονική γνώση για να ε, βοηθήσουμε την προστασία των ζώων στην Ευρώπη. Επίσης, οι χώρες μέλη μας ε, ζητάνε πράγματα, όχι πολύ συχνά. Και τέλος, ακόμα και αν κανείς δεν μας το ζητήσει, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, αναλαμβάνουμε εμείς την πρωτοβουλία για να είμαστε έτοιμοι για μελλοντικέ ερωτήσεις που θα μας έρθουν. Οπότε έχουμε εντολή από τους τέσσερις αυτούς πελάτες, ας το πω έτσι, και τότε ξεκινάει το επιστημονικό μας έργο, ε, εκτιμούμε, αξιολογούμε, δίνουμε επιστημονικές ε, γνωμοδοτήσεις, ε, τις εγκρίνουμε και στη συνέχεια τις δίνουμε στους διαχειριστές κινδύνου. Και ποιος ε, την κάνει αυτή τη δουλειά στην ΕΦΣΑ. Είμαστε κάπου 500 άνθρωποι προσωπικό, αλλά έχουμε 10 επιστημονικά πάνελ με 20 εμπειρογνώμονες από παντού από την Ευρώπη. Είτε πρόκειται για την υγεία των φυτών, είτε πρόκειται για τους γενετικά οργανισμούς, για τις οτροφές, για την προστασία των ζώων, για βιολογικούς κινδύνους, για χημικά, για προσθετικά στα τρόφιμα, συσκευασία κλπ. κλπ. Οπότε πηγαίνουμε από την υγεία των φυτών μέχρι τα τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση εξετάζουμε όλο το σύστημα και κοιτάμε και τους αναδιόμενους κινδύνους. Είναι καθήκον μας να προσπαθούμε να κοιτάμε μπροστά και να σκεφτούμε τι νέοι κίνδυνοι θα προκύψουν εξαιτία τη μετανάστευση, α πούμε, εξαιτία τη καινοτομία στην ε, βιομηχανία τροφίμων. Ε, τι κίνδυνοι θα βρεθούν στο δρόμο μα στο μέλλον και να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτή η προετοιμασία είναι ένα στοιχείο κλειδί θα έλεγα του έργου μας. Και το έχουν υπόψη τους όλα τα πάνελ μας και όλοι στο προσωπικό μας. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι και οι πέντε οργανισμοί εργαζόμαστε μαζί για μία υγεία, ένα πλανήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. You were so Φαίνεται ότι είστε απόλυτα ε, ε, έτοιμοι να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Τελευταία, πριν ε, δώσουμε το λόγο στα μέλη για να λάβουν το λόγο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, εκτελεστικός διευθυντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Είναι χαρά να παρουσιάζω το έργο του Ευρωπαϊκού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος εδώ στην Επιτροπή σας. Φέτος κλείνουμε 25 χρόνια και η βασική δουλειά μας είναι να δίνουμε γνώσεις ε, στους Ευρωπαίους ηθήνοντες ε, για να βελτιώνουν το περιβάλλον και το κλίμα στην Ευρώπη και να ενισχύουν τη συνεισφορά της Ευρώπης στην παγκόσμια προκλήσεις στον τομέα αυτό. Αυτό το οποίο κάναμε τα 25 αυτά χρόνια είναι να παρέχουμε έγκαιρες, αξιόπιστες, στοχευμένες και σχετικές πληροφορίες ε, στους ε, ηθήνοντες, ε, ώστε εσείς και οι υπόλοιποι να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει στοιχείων για το περιβάλλον και το κάνουμε και με την Επιτροπή σας, αλλά και με αρκετές άλλες επιτροπές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεργαζόμαστε με πάνω από 10 υπηρεσίες της Κομισιόν, με προτεραιότητα φυσικά τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τη Γενική Διεύθυνση Κλίματος, αλλά φυσικά συνεργαζόμαστε και ε, στενά με τα κράτη-μέλη. Αυτό το κάνουμε με πολιτικές που αφορούν την ποιότητα των υδάτων, την ποιότητα του αέρα, διαχείριση αποβλήτων, ε, κλιματική αλλαγή, αλλά και συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα υγεία και περιβάλλον. Και έχουμε λοιπόν και συνεργασία με κάποιους από τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ σήμερα. Όλα αυτά γίνονται ε, σε σχέση με παγκόσμια θεματολόγια για το κλίμα, αλλά και με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης πλέον. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό δίκτυο με τις χώρες μέλη. Έχουμε 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 11 επιπλέον χώρες και μαζί με αυτές ε, διαχειριζόμαστε και συγκαλούμε δίκτυα εμπειρογνωμόνων, πάνω από 3.000 δίκτυα που ε, συγκεντρώνουν τους καλύτερους εμπειρογνώμονες για θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία που βελτιώθηκαν στις γνώσεις μας τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι αντιληφθήκαμε ότι τα προβλήματα και οι λύσεις πρέπει να θεωρούνται ως συστήματα, σε επίπεδο συστήματος δηλαδή. Όταν βλέπουμε τις προκλήσεις είναι προφανές ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή κλιματική κρίση αυτή τη στιγμή, αλλά επίσης αντιλαμβανόμαστε όλο ένα και περισσότερο και χαίρομαι γι' αυτό ότι η βιοποικιλότητα συνδέεται άρρηκτα με το κλίμα και αντιστρόφως. Και επίσης εξετάζουμε και ε, την μη βιώσιμη χρήση πόρων και τον αντίκτυπο που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Και τα μηνύματα νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφή. Πρόκειται για μια κατεπίγουσα κατάσταση. Έχουμε ήδη ε, σημεία τα οποία είναι μία αναστρέψιμα και πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Και στο προηγούμενο ε, θέμα συζητήσατε τα συνήθη, ότι δεν αλλάζει τίποτα. Να σας πω ότι όσον αφορά το περιβάλλον δεν υπάρχει πλέον ε, το συζητούμε τα συνήθη. Έχουμε περάσει στον τομέα του ασυνήθιστου και πηγαίνουμε σε αχαρτογράφικα τα νερά. Αυτό σημαίνει ότι οργανώνουμε τις γλώσσες μας... Ε, βάση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων πολιτικής ε, που θα πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένο επίπεδο, σε επίπεδο ενέργειας, σε επίπεδο κινητικότητας και στο σύστημα των τροφίμων. Εάν το μεταφράσω αυτό σε θεματολόγιο πολιτικής, προφανώς ε, το Green Deal, το οποίο εντάσσεται και στις ε, πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της μελλοντική Προέδρου τη Ursula von der Leyen περιλαμβάνει συγκεκριμένε και αυξημένε φιλοδοξίε σε πολιτικό επίπεδο και πρέπει να πω ότι ασχολούμαστε με όλε. Η σύνοψη του θεματολογίου είναι σαν το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών μα ε, ε, από πολλέ πτυχέ. Υπάρχει φυσικά η σχέση με το κλίμα και την ενέργεια. Εκεί είμαστε αρμόδια για παροχή στοιχείων και πληροφοριών για ε, ενέργειες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ασχολούμαστε με τη στρατηγική για τη βιοπικιλότητα και ο στόχος είναι να πάμε στην COP στην Κονίνο που θα έχουμε και ε, μια φιλόδοξη στρατηγική για την ε, βιοπικιλότητα. Για το μη τοξικό περιβάλλον είμαστε τοποθετήριο τον, ε, τις οδηγίες για τις βιομηχανικές εκπομπές και τη ρήπανση. Η βιοοικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, διότι βλέπουμε πάρα πολύ τα θέματα της βιομάζας και τι μπορεί να παρέχει για την ε, κοινωνία και φυσικά υπάρχουν και πολλά ανταλλάγματα και μας αφορά φυσικά και η κυκλική οικονομία και συμμετέχουμε και σε αυτό. Ε, και την πρωτοβουλία για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, η ονοματολογία που έχει δοθεί, ε, συμμετέχουμε σε όλα αυτά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τους περιβαλλοντικούς και τους ε, κλιματικούς στόχους και να τεθούν επιτάπητος. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι συμμετέχουμε πλήρως σε αυτό το θεματολόγιο που έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν την έκθεση IPCP, IPCC και έχουμε και την έκθεση για την βιοπικιλότητα και τα οικοσυστήματα και το πάνελ των πόρων. Συμμετέχουμε σε μεγάλο βαθμό και σε αυτέ τι εργασίε και κάθε πέντε χρόνια η Ευρώπη συγκεντρώνει τι καλύτερε γνώσει τη και αυτό αποκαλείται το SOER, η κατάσταση και η πρόβλεψη ε, των πόρων. Υπάρχει μια τέτοια έκθεση κάθε ε, πέντε χρόνια και η διαφορά με τις άλλες εκθέσεις είναι ότι η δική μας ε, αφορά ρητά το θεματολόγιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ξέρουμε πού βρισκόμαστε και αν δείτε τους στόχους του 2020 για την Ευρώπη, Κατά βάση είμαστε κίτρινο και κόκκινο, υστερούμε στα, όσον αφορά τους στόχους, αλλά έχουμε και γνώσεις οι οποίες μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα φιλόδοξο 2020 και 2050. Αυτή τη στιγμή ε, είναι στη διαδικασία της εκτύπωσης η έκθεση. 4 ε, Δεκεμβρίου θα ε, παρουσιαστεί στο Συμβούλιο εδώ στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος ε, ήδη δεσμεύτηκε ότι θα είναι παρόν. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα υπάρχει παρουσία του Επιτρόπου και της Προεδρίας και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα κάνουμε σε αυτή την έκθεση είναι ότι θα δώσουμε την υφέρπωση ανάλυση για το λόγο ύπαρξης ενός Green Deal για την Ευρώπη και την ευθύνη της Ευρώπης ανά τον κόσμο. Και φυσικά θα δώσουμε στοιχεία για τη δυναμική της μεταβατικής αλλαγής η οποία θα πρέπει να γίνει για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω τα μηνύματα εκεί είναι σαφή. Η, ε, στόχοι και τα όσα έχουμε κερδίσει δεν θα μας οδηγήσουν στο 2020 και το 2050 για το κλίμα. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα όσα κάνουμε, αλλά και με διαφορετικό τρόπο και ότι πρέπει να υπάρχουν ε, αλλαγές, όχι μόνο για τις τρέχουσες πολιτικές, αλλά να έχουμε και πληροφορίες για τα όσα θα χρειαστούμε στο μέλλον και αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς ε, στην υπηρεσία μας. Ε, Φυσικά συνεργαζόμαστε με χαρά μαζί σα, Παραδοσιακά προσκαλούμε εισηγητέ αρμόδιους για θέματα να έρθουν στην υπηρεσία για να του δώσουμε τι καλύτερε ε, δυνατέ πληροφορίε. Υπάρχει πρόσβαση σε δίκτυα επιστημόνων που ε, μπορεί να είναι χρήσιμα για το δίκτυο αυτό και ε, θα ήθελα να τονίσω ότι όλο και περισσότερο συνεργαζόμαστε με του συναδέλφου εδώ για να έχουμε μια προοπτική, ένας πλανήτης, μια υγεία και πάντα να λαμβάνεται αυτή η υπόψη. Ε, ο συνάδελφος από την ΕΦΣΕ είπε ότι βασίζεται στη συζητήση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να έχουμε περαιτέρω θέσει εργασίας και πόρους για τη δική του την υπηρεσία. Μακάρι να μπορούσα να πω και εγώ το ίδιο. Εμείς ε, δυστυχώς είμαστε στην κατηγορία των υπηρεσιών που έχει περικοπές ε, στους πόρους που είναι και κάπως παράδοξο δεδομένων των προτεραιοτήτων που έχουμε για το μέλλον στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και κάνω έκκληση το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να διαδραματίζει τον πολύ θετικό ρόλο του και να δεσμευτεί για την κατάλληλη διάθεση πόρων σε υπηρεσίες οι οποίες κάνουν την καθημερινή δουλειά που χρειάζεται για να ε, εκπληρούν τις υποσχέσεις προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μου άρεσε αυτό που είπατε για τις ασυνήθιστες και τα αρθαχαρτογράφικα τα νορά. Ε, έχουμε πάει στο σωστό πλαίσιο. Πάμε στον αρμόδιο με την ΕΜΒΗ. Θα ξεκινήσουμε με το Μάρτιν Χότζινγκς από το Ρινιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Νομίζω ότι η υπηρεσία για τα χημικά είναι μια υπηρεσία που έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για τη διαχείριση των χημικών και την προπτική της βιομηχανίας χημικών, αλλά ε, προστατεύει και την υγεία και το περιβάλλον αφενός και εξασφαλίζει και την ε, αντικατάσταση ε, κάποιων ουσιών, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μας είπατε στην παρουσίαση, την ε, πολύ σημαντική διαδικασία αδειοδότησης και της αντικατάστασης ε, κάποιων επικίνδυνων χημικών. Και θεωρώ ότι αυτό δεν αφορά μόνο την υγεία και το περιβάλλον, αλλά θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικός μοχλός καινοτομία, διότι εκεί δημιουργείται ο μηχανισμός, ο οποίος ε, ουσιαστικά δίνει κίνητρα για να δώσουμε ευκαιρία για τις επιχειρήσεις για να επενδύσουν στο μέλλον, γιατί ξέρουν ότι θα υπάρχει μια αγορά αν υπάρχει, για παράδειγμα, ε, μια ασφαλής εναλλακτική λύση για ένα χημικό καρκινογόνο. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς ε, θα δούμε τα θέματα των χημικών από κοινού, γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση ε, είναι ως εξής. Υπάρχει μια σειρά από άλλα νομοθετήματα και τα βλέπουμε ανά σκέλος. Για παράδειγμα, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ή νομοθεσία για τα καλλιντικά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που πρέπει να κάνουμε λοιπόν και το Green Deal είναι πολύ σημαντική συνιστόσα, αλλά επίσης αυτό το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό είναι η, υπηρεσία των χημικών να έχει κατάλληλους πόρους ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ε, διότι χωρίς ε, ισχυρούς και ποιοτικού ε, ρυθμιστές δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική αγορά νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αλλά δεν εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Μποναφέ για το γεγονός ότι δεν παρεμπιρίσκεται στη σημερινή συνεδρίαση, αλλά αυτό οφείλεται σε κάποιες περιστάσεις που δεν μπορούσε να προβλέψει. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας σήμερα εδώ, ε, γιατί μας βοηθάτε να αντιληφθούμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος της ΕΦΣΑ ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ε, τροφίμων. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία η οποία συνήφθη ε, νωρίτερα φέτο, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ευρύτερη νομοθεσία κατά τρόφιμα, αυτά θα ε, κληθεί να αναλάβει πολύ διαφορετικά καθήκοντα μέσα στα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια αλλά και την εμπιστευτικότητα. Ε, οι κανόνες δηλαδή σε αυτή τη φάση, αυτή τη σήμερον ημέρα, ανάλογα με τον κάθε τομέα, διαφέρουν. Ενώ με τους, νέου κανόν, με τους νέους κανόνες οποιαδήποτε αίτηση για διοδότηση θα δημοσιεύεται χωρίς καμία καθυστέρηση μόλις θα θεωρείται ως έγκυρη ε, μια αίτηση. Ταυτόχρονα έφασα θα πρέπει να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων ε, για ε, τις μελέτες οι οποίες θα συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση για την αδειοδότηση με αυτόν τον τρόπο η ΕΦΣΑ θα μπορεί να παρέχει συμβουλές ε, στον κάθε Οπότε θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω ποια μέτρα λαμβάνει η ΕΦΣΑ προκειμένου να αλλάξει την ιστορική της οργανώση έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα νέα καθήκοντα και ένα Δεύτερο ερώτημα είναι, ε, θεωρείτε πως ο τρέχον προπολογισμό θα είναι επαρκής έτσι ώστε να μπορέσει η ΕΦΣΑ να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες ευθύνες που θα αναλάβει. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε Ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, είναι, δεν έχει καταφέρει από τα μέσα της δεκαετίας του 90 να μειώσει την ε, χρήση των ε, φυτοφαρμάκων. Ε, και έχετε κάποιους δείκτες σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα από την χρήση των φυτοφαρμάκων, γιατί αυτό αποτελεί βέβαια κάτι ε, το πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Λόγω λοιπόν εναρμονισμένοι δείκτε που έχουν προταθεί τώρα είναι κατάλληλοι ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε αυτό τον αντίκτυπο δηλαδή ε, της χρήσης των ε, αυτοφαρμάκων. Επόμενο μιλήτρια. Ναι. Από ό,τι άκουσα, ο Οργανισμός σε Περιβάλλοντος υποβάλλει μία έκθεση ανά πέντε χρόνια, παρέχοντας μία πλήρη επισκόπηση ως προς τα όσα συμβαίνουν. Αυτή η περίοδος ε, των πέντε ετών είναι ίδια με την περίοδο της βουλευτικής μας ε, θητείας. Ουσιαστικά την, έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή, να διαβάζουμε μία μόνο έκθεση αναθετία. Μήπω θα μπορούσε να υπάρχει μια ενδιάμεση έκθεση, για παράδειγμα, έτσι ώστε να είμαστε σε, σε θέση να παρακολουθούμε καλύτερα τι εξελίξει. Ευχαριστώ, λέει ο Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Κυρία Λιπονόβακα από το ΕΛΚ. Και συνέχεια βέβαια όταν θα ακούσουμε και αυτές τις ερωτήσεις θα έχουν τη δυνατότητα και οι εκπρόσωποι των οργανισμών να απαντήσουν. Κυρία Νόβακ λοιπόν. Ναι. Ε, καταρχήν να σας πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη για, τις, ε, για την ενημέρωση ε, που έλαβα σήμερα σε σχέση με αυτούς τους οργανισμούς της Ένωσης και το πώς υποστηρίζουν την προετοιμασία της νομοθεσίας που παράγουμε. Η Επιτροπή μας βέβαια είναι μια επιτροπή που καλύπτει μεγάλο φάσμα ζητημάτων και εγώ ως ε, νέο μέλος της ε, συχνά διαρωτώ με ε, ποιον θα πρέπει να έρθω σε επαφή, σε ποιον θα πρέπει να βασιστώ όταν αντιμετωπίζουμε μια σειρά από διαφορετικά ζητήματα εδώ, όταν τα εξετάζουμε. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και τα διάφορα λόμπι, τα οποία βέβαια κάνουν την δική του δουλειά και ασκούν τι δικέ του επίεσει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα λοιπόν έχω ένα επαναπαυθεί λίγο γιατί βλέπω με ποιον τρόπο εργάζεστε. Αλλά εκείνο που διαρωτώ είναι Ποια είναι η βάση για την νομοθεσία μας. Ε? Σε αυτή τη διαδικασία ε, συμμετέχουν δηλαδή μόνο αξιωματούχοι, αν θέλετε, από διάφορε υπηρεσίε ή και εμπειρογνώμονε. Ε? Είχα αυτό το ερώτημα και διαπιστώνω με χαρά μου ότι πράγματι οι διάφοροι οργανισμοί σα έχουν μεγάλο έχουν υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνη. Γιατί πράγματι τέτοιο είδου προετοιμασία θα πρέπει να βασίζεται σε, σε όσο το δυνατόν περισσότερη εμπειρογνωμοσύνη. Είναι δηλαδή αλήθεια ότι το Κοινοβούλιο βασισμένο σε τέτοιου είδους ε, εμπειρογνωμοσύνη μπορεί στη συνέχεια να λάβει πολιτικέ ε, αποφάσεις. Δηλαδή, ο πολιτικό χαρακτήρα μια απόφαση να βασίζεται και να ευθυγραμμίζεται με την ε, εμπειρογνωμοσύνη. Βέβαια, συχνά τέτοιου είδου ζητήματα αποκτούν και ένα πολιτικό χαρακτήρα, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω σε αυτό. Απλώ χαίρομαι με αυτές τις παρουσιάσεις που άκουσα σήμερα και γνωρίζω τώρα με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω όταν θα χρειάζομαι πιο εξειδικευμένη ενημέρωση, όταν θα χρειάζομαι εμπειρογνώμοσύνη για να τοποθετηθώ σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη που μας παρέχετε και βέβαια ελπίζω όταν κάνετε και εσείς ασκείτε τα δικά σας καθήκοντα, λαμβάνετε υπόψη σας ε, ε, το ρόλο του Κοινοβουλίου. Στον επόμενο γύρο είχα ζητήσει εγώ το λόγο, όχι τώρα. Uh, It's this one for you. So, Anya Azekamp for the GUE. Yes. Η Άνια Αζεκάμπ για την ΓΚΟΕ e τώρα. Ναι, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον ε, ε, κύριο Χάντσεν από τον Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και μετά ε, προς την Χθε λοιπόν είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσκεψη σε ό,τι αφορά του ενδοκρινικού διαταράκτε. Και βέβαια η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματο των ενδοκρινικών διαταρακτών αποτελεί ένα από τα βασικά τώρα προβλήματα αυτή τη γενιά αλλά και των επόμενων γενιών. Και η πρόοδο που επιτελείται εδώ είναι πολύ αρκή. Πώ μπορούμε λοιπόν να επιτυχίνουμε τη διαδικασία αναγνώριση λοιπόν και απαγόρευση όλων αυτών των ενδοκρινικών διαταρακτών από όλα τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μα ζωή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε ενδεχομένω μια ε, προσέγγιση ομαδοποίηση σε ό,τι αφορά δηλαδή οι ουσίε με τι παρόμοιε ιδιότητε έτσι ώστε να αποφύγουμε περιπτώσει ε, υποκατάσταση ε, και να μην έχουμε περιπτώσει όπω για παράδειγμα τη υποκατάσταση του bisphenol A με το bisphenol C όπω έγινε. Επίση, ακούσαμε ότι ζητήσατε περισσότερου πόρου από τη δική σα πλευρά και υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. Αλλά μήπω χρειάζεστε και παραπάνω ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να είστε σε θέση να αντιδράτε ταχύτερα στι νέε προκλήσει. Τώρα, το ερώτημά μου προ την ε, Ασφάλεια Τροφίμων, τον μου. ε, Μα ανησυχούν πολύ οι περίοδοι που βλέπουμε και οι παρατάσει που δίνονται σε αυτέ τι περιόδου για την έγκριση των φυτοφαρμάκων. Δηλαδή, βλέπουμε από το 2003 ε, και μετά να υπάρχει παράταση που δίνονται μέχρι και για πέντε συναπτά έτη επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Και αυτό ισχύει και για ε, φυτοφάρμακα τα οποία μπορούν να είναι και ε, καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα, να έχουν αρνητικέ επιπτώσεις στην αναπαραγωγή και να είναι και ενδοκτηνική Διαταράκτε Βέβαια υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσει οι οποίε προκύπτουν σε επίπεδο αξιολόγηση από πλευρά των κρατών μελών, αλλά και εσεί κάνετε τέτοιε καθυστερήσει και θα θέλαμε να μα πείτε το γιατί και τι μπορεί να γίνει για να τι αποφύγουμε. Συγκεκριμένα μπορείτε να μα εξηγήσετε γιατί δεν έχετε ακόμα δημοσιεύσει την δική σα νομοδότηση σε ό,τι αφορά το Μάνκο ΣΕΠ, γιατί η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018. Και η Επιτροπή αξιολόγηση του Κινδύνου από την πλευρά ε, του ΕΚΑ ε, έχει πράγματι τοξικές επιπτώσεις για την αναπαραγωγή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να απαγορευτεί άμεσα. Ε, και γιατί ακόμα εσείς δεν έχετε προετοιμάσει τη δική σας γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος για το ίσια τώρα κύριο Σόκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επικεφαλή των διαφόρων οργανισμών για τις παρουσιάσεις τους. Εγώ ένα σύντομο να σχόλιο να κάνω από τη δική μου πλευρά. Η δημόσια διαβούλευση αποτελεί ένα πολύ ισχυρό δημοκρατικό εργαλείο και αποτελεί και επίση ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο για να συλλέξετε δεδομένα σε ό,τι αφορά κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα αλλά και επιστημονικά, επιστημονικέ επιτυχίε. Άρα λοιπόν η μόνη κριτική που μπορώ εγώ να ασκήσω σε αυτό το, το εργαλείο τη δημόσια διαβούλευση είναι το γεγονό ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερε οργανώσει λόμπι αλλά και οι μεγαλύτερου μεγέθου, αν θέλετε, ε, με κυβερνητικέ οργανώσει έχουν πρόσβαση σε αυτό. Ενώ αντιθέτω οι μικρότερε οντότητε, οι μικρότεροι οργανισμοί έχουν ε, δυσκολία στο να έχουν πρόσβαση και να τοποθετηθούν στο πλαίσιο αυτής της δημόσιας διαβούλευση. Αυτό βέβαια οφείλεται κυρίω στην ε, ενημέρωση για την επίγνωση ότι υπάρχει μια τέτοια δημόσια διαβούλευση, αλλά γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα πρέπει να την ε, τονίζουμε ω διαδικασία όλο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε να συλλέγουμε και όσο το δυνατόν περισσότερα σχόλια. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Μάργαρετ και τώρα για του ε, πράσινου. Ναι, ε, απευθύνομαι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο ε, και να πω ότι πραγματικά είναι δραματικό το γεγονό ότι έχει προβλεφθεί περικοπή του προπολογισμού του. Αλλά έχετε προτείνει κάτι σε ό,τι αφορά την στρατηγική για τα πλαστικά. Από τη δική σα πλευρά, ίσω να μην γνωρίζω κάτι το οποίο έχετε δημοσιεύσει, γιατί θυμάμαι ότι είχατε πει από, από κάποια χρόνια ότι θα, τοποθε, θα ε, υπήρχε μια στρατηγική από τη δική σα πλευρά για τα πλαστικά, ανεξαρτήτω δηλαδή τη στρατηγική που θα θετούσε εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γνωρίζουμε ότι σα έχουν ασκηθεί πιέσει προ αυτή την κατεύθυνση και στο πλαίσιο γενικότερα τη πολιτική σε ό,τι αφορά τα ε, απορρίμματα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε και την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη από τη δική σα πλευρά, από τον Οργανισμό Περιβάλλοντο, σε σχέση με τη χρήση των πλακτικών, για να έχουμε και ένα ακόμα ε, επιχείρημα ε, προκειμένου να ταχθούμε υπέρ τη ενίσχυση τη αύξηση του προπολογισμού σα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ένα ακόμα ομιλητή και μετά και εγώ θα θέσω τα δικά μου ερωτήματα. Α, όχι, βλέπω και άλλου ομιλητέ που θέλουν να πάρουν το λόγο, ωραία. Ευχαριστώ. Περισσότερα από ένα ερώτημα θα ήθελα να θέσω. Καταρχήν το πρώτο μου ερώτημα αφορά το ΝΕΦΣΑ γιατί εδώ έχω συμπογράψει μια επιστολή που σας αποστήλαμε και για την οποία δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί γνωρίζουμε πως το έλυσε. δεν θεωρείται ως ιδιωτικός οργανισμός από την πλευρά ε, του ΕΦΣΑ, παρότι ο, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας τη θεωρεί ως ιδιωτικό φορέα. Οπότε ποιο ρόλο θα παίξουν αυτά τα μέλη αυτού του λόμπι, αυτή η εκπρόσωπη λόμπι. Γιατί αν εσεί του θεωρήσατε στο μέλλον ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, αυτό θα με ανησυχούσε. Το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να σας ε, θέσω είναι το εξή. Στη διαφάνειά σας εδώ μας παρουσιάσατε ε, το ζήτημα τη ενημέρωση των κινδύνων και ακούσαμε από την πλευρά του οργανισμού περιβάλλοντος, ε, κάποια περισσότερο σε ό,τι αφορά την κρίση σε σχέση με τη βιοπικιλότητα. Πώς λοιπόν θα λάβετε υπόψη σας αυτή την πτυχή σε ό,τι αφορά ε, δυνητικά ε, σενάρια, δηλαδή υποβάθμιση του εδάφους ακριβώς λόγω της κρίσης της βιοπικιλότητας. Πώς αυτό δηλαδή θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην παραγωγή τροφίμων μα ή στον τρόπο με τον, τις γεωργικές μας δραστηριότητε. Το έχετε εξετάσει αυτό ή για παράδειγμα έχετε εξετάσει το ποιε θα ήταν οι επιπτώσει, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά ε, την περισσότερη διάδοση των νόσων, επειδή δεν υπάρχουν και οι θηρευτέ, δηλαδή τα ζώα τα οποία κυνηγούν. Μετά, σε ό,τι αφορά τον οργασμό ε, ε, φαρμάκων, μήπω θα ήταν πιο δίκαιο να αυξήσετε τα τέλη τον που πρέπει να καταβάλουν επιχειρήσεις εκείνες, ειδικότερα εκείνες που έχουν υποβάλει ε, φακέλους οι οποίοι δεν ήταν πλήρες, αντί να ζητείτε απλά αύξηση του προπολογισμού από πλευρά της Ένωσης. Ευχαριστώ. Φοβάμαι ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη διάκριση. Στην Κροατία, στη χώρα μου, συχνά υπάρχουν τρόφιμα κακής ποιότητας που κυκλοφορούν στην αγαρά μας. Είναι γνωστές περιπτώσεις γαλακτοκομικών προϊόντων που δεν μπορούν να απολυθούν σε άλλες χώρες, αλλά στην Κροατία απολούνται. Βλέπουμε πολλές φορές επίσης σκάνδαλα για τέτοια προϊόντα. Έχει γίνει μεγάλη ιστορία με αυτά με την ουτέλα. Υπάρχει διάκριση σε βάρο μας. Στη Γερμανία η νουτέλα που πλειόταν εκεί ήταν πολύ καλύτερης ποιότητας από αυτήν που είχαμε εμεί στην ε, χώρα μας. Οπότε θέλω να ρωτήσω την Εύσα, τι μέτρα λαμβάνονται για να σταματήσει αυτή η ανισότητα και αυτές οι διακρίσεις που γίνονται. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλες οι χώρες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια ποιότητα προϊόντων και καμιά χώρα να μην θεωρείται ως νεκέ των άλλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς έχει ζητήσει το λόγο. Όχι. Λοιπόν, η δικιά μου ερώτηση τώρα. Προς την ΕΚΑ και την ΕΦΣΑ για το εφέ κοκτέιλ. Γιατί βλέπετε δεν είναι κατακαιρματισμένο το ανθρώπινο σώμα. Εσείς είσαστε διάφορες ε, οργανώσεις. Εμείς Είμαστε ένας οργανισμός ε, ενωπημένος. Οπότε το θέμα δεν είναι να κοιτάμε τα πράγματα μόριο-μόριο ή ουσία, η ουσία ο καθένας ε, στο πεδίο του, γιατί στο τέλος η υγεία είναι μία υγεία. Οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται και απαιτείται από σας τεχνικά, αλλά ίσως και από πολιτική άποψη, να το δείτε αυτό που αποτελεί ένα νέο όριο που πρέπει να ξεπεράσουμε αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ε, χημικών και της υγείας. Λοιπόν, τώρα, θα σας ζητήσω να απαντήσετε συγκεκριμένα στις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις που ακούστηκαν. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και μετά με τη σειρά. Ωραία, ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις ερώτηση για την έκθεση κάθε πέντε χρόνια. Εμείς κάνουμε κάπου 40 εκθέσεις κάθε χρόνο. Φυγραμμιζόμαστε απόλυτα στην ε, παράδοση των οργανισμών που ασχολούνται με διάφορα θέματα. Ε, κάθε πέντε χρόνια συγκεντρώνετε την γνώση σας και την παρουσιάζετε όπως το κάνει και το IPCC και UNEP και διάφορες διεθνείς οργανώσεις. Αυτή είναι η παράδοση που ακολουθούμε εμείς και αναφέρεται και στον κανονισμό μας. Αυτό κάνουμε. Ε, κάνουμε αιτήσια έκθεση για την ποιότητα του αέρα, των υδάτων, για τη βιοπικιλότητα κλπ. κλπ. Αυτά τα κάνουμε σε αιτήσια βάση. Επίσης έχουμε πλατφόρμες οι οποίες συνεχώς ενημερώνουν τα δεδομένα. Το σύστημα για την ποιότητα των υδάτων, για παράδειγμα για τη βιοπικιλότητα ή για το κλίμα ενημερώνονται συνεχώς με τη νέα γνώση που αποκτάμε. Και έχουμε επίσης επενδύσει και πολύ σε έναν διαφορετικό τρόπο για να φτάνουμε στους πολίτες. Που σημαίνει ότι μερικές φορές ώρα την ώρα ενημερώνουμε με τα νέα δεδομένα και μπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε πόλη 10.000 ή παραπάνω να πατήσετε στο χάρτη πάνω σε αυτή τη χώρα και να δείτε ποια είναι η ποιότητα του αέρα τη συγκεκριμένη ώρα. Γίνεται αυτή η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο θα μας βοηθούσε είναι οι επενδύσεις στο Κοπέρνικους. Έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στο σύστημα αυτό παρατήρησης του πλανήτη και τα δεδομένα τα οποία μας προσφέρει είναι πολύ πιο καλά και έρχονται πολύ πιο γρήγορα από άλλες αιτήσεις παρατηρήσεις που γίνονται από κάποιες χώρες και μας αποστέλλονται. Κάνουμε λοιπόν πολύ περισσότερο από ότι μία έκθεση κάθε πέντε χρόνια που είπατε. Τώρα, για τη βιοπικιλότητα και την κρίση βιοπικιλότητας σε σχέση με τη Γεωργία. Δεν έχει απευθεία σχέση με μας, αλλά έχουμε την έκθεση για την βιοπικιλότητα και η κυριότερη πίεση στη βιοπικιλότητα στην Ευρώπη είναι το σημερινό αγροτικό σύστημα. Το άλλο είναι ο κατακαιρματισμός της γης και το τρίτο είναι η ρήπανση. Και όλα αυτά ακούστηκαν στις ερωτήσεις σας. Η κατάσταση λοιπόν είναι ότι το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε ότι μέχρι το 2010 θα σταματήσει την απώλεια βιοπικιλότητας. Μετά είπε το 2020 ούτε και αυτό θα γίνει. Τώρα ε, ε, θα διονυστεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να πούμε πια τι θα κάνουμε το 2030. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο οδηγεί στην απώλεια βιοπικιλότητας πρέπει να αντιμετωπιστεί και το κυριότερο είναι τα αγροτικά συστήματα και οι πολιτικές που επιδοτούν αυτά τα συστήματα. Και αυτό το αναφέρουμε σε πολλές από τις εκθέσεις μας. Αυτέ είναι νομίζω κυρίω οι ερωτήσει οι οποίε απευθύνθηκαν σε εμά. Α, για τα πλαστικά, για τη στρατηγική για τα πλαστικά επίση ρωτήσατε. Λοιπόν, όπω γνωρίζετε δεν είμαστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχουμε εμεί το δικαίωμα πρωτοβουλία. Εμεί συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των, πλακτικών, των πλαστικών με πολλού και διάφορου τρόπου. Πρώτα απ' όλα για τα χημικά και την υγεία. Στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το έργο. Δεύτερον, μη τοξικό περιβάλλον που ενσωματώθηκε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια πρωτοβουλία πολιτικής. Μένει τώρα στην Επιτροπή να δει τι θα κάνει. Έπειτα, το θέμα των αποβλήτων. Με τα πλαστικά βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει να διαχειριστεί τα δικά της πλαστικά. Η Κίνα και άλλες χώρες δεν δέχονται πια τα δικά μας απόβλητα. Οπότε δουλεύουμε στην κυκλική οικονομία και για τα πλαστικά, κάτι το οποίο όμως είναι δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο το πλαστικό υλικό να χρησιμοποιηθεί στην κυκλική οικονομία. Είναι ένα υλικό το οποίο δεν ε, διατηρεί την ε, αξία του και δεν μπορεί να παραχρησιμοποιηθεί στην κυκλική οικονομία. Οπότε προσπαθούμε και εμείς ε, να βοηθήσουμε με την στρατηγική για τα πλαστικά όσο μπορούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις που μας κάνετε. Θα απαντήσω κι εγώ όσο μπορώ καλύτερα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τη νέα ρύθμιση για τη διαφάνεια. Τι θα αλλάξει, όπως ίσως γνωρίζετε, ο νέος κανονισμός για τη διαφάνεια αποτελείται από τέσσερις επιλώνες. Διαφάνεια, ποιότητα μελετών που χρησιμοποιούμε, ποιότητα δεδομένων δηλαδή, ε, διακυβέρνηση της ΕΦΣΑ και τέταρτον επικοινωνία. Όσον αφορά τη διαφάνεια λοιπόν, εμείς όπως προβλέπετε στην νομοθεσία από τον Μάρτιο του 2021, τότε δηλαδή που πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία, θα δημοσιεύσουμε όλα τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τις αξιολογήσεις μας αμέσως μετά από τη στιγμή που θα έχουν υποβληθεί οι αιτήσει. Θα αντελέξουμε και μετά από λίγε εβδομάδε θα δημοσιεύσουμε όλα τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση κινδύνου που κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προ τα μπρο. Όχι μόνο για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού, αλλά και επιστημονικά μιλώντα. Γιατί άλλοι ερευνητέ θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα με τι δικέ του μεθοδολογίε, με τα δικά του στατιστικά και τα δικά του πρότυπα και ίσω μπορεί να βρούνε κάποια ε, πράγματα τα οποία εμείς να μην τα βλέπουμε. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό και από ό,τι ξέρουμε κανείς δεν το έχει αυτό στον πλανήτη. Η Ευρώπη εδώ είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη διαφάνεια και ε, με το δικιά μας πολιτική ε, του να είμαστε ανοιχτοί δηλαδή, πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε πολύ. Τώρα, όσον αφορά την ποιότητα των μελετών, θα έχουμε ένα μητρό μελετών, οπότε και ο κλάδος και τα εργαστήρια τα οποία εκπονούν τις μελέτες θα τις κοινοποιούν πριν, τις, πριν γίνουν οι αιτήσει, οπότε δεν θα χάνετε καμία ε, έκθεση στο δρόμο. Τώρα, θα αλλάξει επίσης και η διακυβέρνησή μας. Έχουμε τώρα ένα διοικητικό συμβούλιο με τις χώρες μέλη, με 14 άτομα που έχουμε με ανοιχτό διαγωνισμό αλλά μετά οι χώρε μέλη, το κοινοβούλιο, η κοινωνία των πολιτών θα εκπροσωπούνται όπως συμβαίνει με όλες ουσιαστικά με όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και όσον αφορά την επικοινωνία μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει μια εκτελεστική πράξη για ένα σχέδιο κοινών ανακοινώσεων όπου θα υπάρχει μια κοινή προσέγγιση. Κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ θετικό κατά τη γνώμη μας γιατί στην ε, ανακοίνωση των κινδύνων μερικές φορές μηνύματα που δεν ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους μπερδεύουν τον κόσμο. Το 2017, για παράδειγμα, υπήρξαν διαφορετικά μηνύματα που έφτασαν προς τον κόσμο και μπερδεύτηκε ο κόσμος. Τώρα φτάνει ο προπολογισμό, ρωτήσατε. Για τα νέα καθήκοντα, αν έχουμε τον προπολογισμό που προβλέπετε, ναι. Αλλά για τις ελλείψεις ε, στα τακτικά καθήκοντα της ΕΦΣΑ, για παράδειγμα και τα φυτοφάρμακα, δεν θα έχουμε παραπάνω χρήματα. Παραπάνω χρήματα είναι για τη διαφάνεια, για την επικοινωνία, για την ποιότητα ε, των εκθέσεων ε, και τη διακυβέρνηση, για τα νέα μας καθήκοντα δηλαδή. Και καλό είναι αυτό. Αλλά Έχουμε ελλείψεις για τα φυτοφάρμακα για παράδειγμα. Έχουμε κάπου 60 ανθρώπους προσωπικό γι' αυτό. Και στο αντίστοιχο ε, των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν 1.100 ε, περίπου. Στον Καναδά επίσης που είναι μια μεγάλη χώρα από πλευράς επικράτειας αλλά είναι πολύ λιγότερος ο πληθυσμός έχουν ε, επίσης πολύ περισσότερους. Οπότε όταν ε, βλέπουμε την ευρωπαϊκή προοπτική και τι δίνει για τα φυτοφάρμακα, εκεί δυσκολευόμαστε. Και θα επανέλθω αργότερα, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τον Ευρωβουλευτή Νόβακ που αναγνωρίζει ότι όντως είναι ανεξάρτητη η υπηρεσία μας. Πρέπει ο κόσμος να το καταλαβαίνει ότι μπορεί να μας εμπιστεύετε Οι οργανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν από εσά, από τον νομοθέτη, απλώς και μόνο για να εξυπηρετήσουν το συμφέρον του κοινού. Τίποτα άλλο. 100% πληρωνόμαστε από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, όχι από τη βιομηχανία. Το μόνο μας καθήκον και μέλημα είναι η προστασία της υγείας του κόσμου. Μας κατηγορούν μερικές φορές να μην είμαστε αρκετά ε, ανοιχτή, με διαφάνεια κτλ. για να σας πείσουμε και να πείσουμε και το κοινό. Κοιτάξτε, ακόμα κι αν δεν μ' αρέσει ε, το αποτέλεσμα για την πολιτική μου, πρέπει να σκέφτεται κανείς, παρόλα αυτά μπορώ να εμπιστευτώ τα δεδομένα. Η νομική σαφήνεια επίσης είναι πολύ σημαντικό για το τι επιτρέπεται και τι όχι να δημοσιευθεί και οι πόροι που δίνονται γι' αυτό. Τώρα για το τελευταίο που με ρωτήσατε, ε, γίνονται συναντήσεις. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω πού βρισκόμαστε, αλλά θα σας ενημερώσω αργότερα. Για τις καθυστερήσεις, ναι, πρέπει να πούμε ότι οι εκθέσεις, τα σχέδια αξιολογήσεων, δηλαδή δεν είναι πάντα της ποιότητας που θα θέλαμε. Γι' αυτό και έχουμε μια διαδικασία αξιολόγηση μεταξύ ομολόγων, ώστε να αξιολογούνται και από τις χώρες μέλη και στο τέλος όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης να είναι του ίδιου επίπεδου. Τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε ένα δίκτυο ε, για τα φυτοφάρμακα με τις χώρες μέλη, με την Επιτροπή για να βελτιώσουμε τη διαδικασία και να την επιταχύνουμε. Αλλά μην κοροδευόμαστε. Έχουμε περιορισμένους πόρους όσον αφορά τα φυτοφάρμακα. Δεν θα μπορέσουμε να διπλασιάσουμε την ταχύτητά μας εκτός αν μπορούμε να έχουμε περισσότερους πόρους. Επίσης, για τη σύγκρουση συμφερόντων με ρωτήσατε. Νομίζω ότι μπορώ να πω με περηφάνεια ότι με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ΕΦΣΑ έχει μια πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με την οποία ο Όμπουτσμαν είπε ότι θα μπορούσαν άλλοι να παραδειγματιστούν από τη ρύθμιση της ΕΦΣΑ. Οπότε έχουμε μια πολύ αυστηρή πολιτική και σας διαβεβαιώ ότι ότι για την περίπτωση της ΕΦΣΑ κατά πόσο θεωρείται ε, ιδιωτικό ή όχι οργανισμό είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε εξετάσει και όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων έχουμε καταλήξει συμπεράσματα. Όταν πρόκειται για τα φυτοφάρμακα, επανέρχομαι σε αυτό, ε, έχει να κάνει με τα χημικά ε, στο έδαφος. Χρησιμοποιούμε τα καλύτερα πρότυπα που διαθέτουμε, αλλά πρόκειται για μία πρόβλεψη. Και μετά όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα υλικά, τότε ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις επί του εδάφους και επί των διαφόρων οργανισμών. Η, ειδική δική σας επιτροπή πρότεινε ότι πρέπει να έχουμε ε, μία έκθεση συνολική για τα φυτοφάρμακα στο περιβάλλον. Εμείς ξέρουμε τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στον άνθρωπο, είναι το καλύτερο σύστημα που έχουμε για τις καθημερινές επιπτώσεις. 80.000 δείγματα έχουμε για τα φυτοφάρμακα και κατά πόσο συμμορφώνονται ή όχι στις ε, ρυθμίσεις. Αλλά όσον αφορά τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον, εδώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Για την ποιότητα τώρα των τροφίμων, για την Κροατία. Για την ποιότητα των τροφίμων δεν έχω αρμοδιότητα εγώ να μιλήσω, γιατί δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Εμείς ε, ασχολούμαστε με την ασφάλεια των τροφίμων όταν αυτά μπαίνουν στην αγορά. Αλλά όταν είναι στην αγορά, ως ασφαλή τρόφιμα, μετά υπάρχει διαφοροποίηση ίσως στην ποιότητα, αν είναι οργανικά ή όχι, τη μάρκα είναι το προϊόν κτλ. Εκεί υπάρχει διαφοροποίηση στην ποιότητα. Αλλά αυτό το εξετάζουν οι χώρες μέλη οι αρμόδιες αρχές των χωρών μελών και όχι ΕΦΣΑ. Για το εφέ κοκτέιλ, θα δώσω το λόγο βέβαια και στο συνάδελφο γι' αυτό. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο οργανισμός μας ε, εκτίθεται σε συνδυασμό ε, ουσιών. Το 2020 την Άνοιξη θα έχουμε τις πρώτες εκθέσεις για τις συνδυασμένε επιπτώσεις των ε, φυτοφαρμάκων επί του νευρικού συστήματος ε, και όχι μόνο. Για 7 χρόνια ασχολούμαστε. Ξέρω, κράτησε πολύ. Θα έπρεπε να είμαστε πιο γρήγοροι. Έχουμε δύο συστήματα. Εμείς κοιτάμε τα φυτοφάρμακα, όχι τα πρόσθετα στα τρόφιμα ή κάτι άλλο. Δεν έχουμε όλη την γνώση πως τα χημικά δηλαδή ε, λειτουργούν ως καταλύτες για να προκαλέσουν κάποιες αντιδράσεις στον οργανισμό. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στην ΕΚΑ και την ΕΦΣΑ, αλλά και των Αμερικανικών υπηρεσιών που έχουν επενδύσει εκατομμύρια σε χημικά μείγματα. Οπότε πρέπει να συνεργαζόμαστε και με τους συναδέρφους από τις ΗΠΑ. Θα συνεχίσουμε το έργο μας για να καλύψουμε και τα επόμενα όργανα είναι μια δουλειά που συνεχίζεται. Θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, ναι, θα μπορούσαν, αλλά... Συμφωνούμε όλοι ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Αν είχαμε περισσότερους πόρους θα κάναμε περισσότερο. Είναι μια έκκληση και προς τους νομοθέτες μήπως κάτι μπορεί να γίνει για να στηριχθεί περισσότερο το έργο μας στην επιστημονική του βάση. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω και εγώ τη σκητάλη από τον Μπέρναρτ και θα πω και δύο πράγματα ακόμα για το εφέ κοκτέιλ, ε, την... Ε, τα μείγματα ουσιών, αλλά να ξεκινήσω με την κυρία Νόβακ και την δική της την παρέμβαση και μετά θα περάσω στα πιο επιστημονικά τεχνικά ζητήματα και τα μείγματα και μετά θα τελειώσω με τη χρηματοδότηση, τα τέλη, τους πόρους κτλ. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα ναι για να ενισχύσω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Εμείς ως υπηρεσία είναι στην εντολή μας ε, να ε, σας υπηρετούμε και φυσικά αυτό επιθυμούμε με ιδιαίτερη προθυμία, ιδίως ε, όταν συζητάτε νομοθετικές προτάσεις που περιλαμβάνουν, περιλαμβάνουν προσθήκη, αλλαγή ε, ή ε, μετατροπή ε, καθηκόντων που αφορά όχι μόνο συζητήσεις πολιτικής αλλά και πόρους, χρονοδιαγράμματα, κατά πόσον είναι εφικτό κάτι, έχει κάποια σκοπιμότητα κλπ. Πολύ ευχαρίστω να συμμετέχουμε σε όλα αυτά. Όσον αφορά τα θέματα ουσίας, να ξεκινήσω με τη δημόσια διαβούλευση, όπου πράγματι Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση. Είναι μεγάλη πρόκληση σε σχέση με το πώς μπορούμε να επιλέξουμε σχόλια, ιδέες και προτάσεις από τους Ευρωπαίους πολίτες ε, να δούμε και τις κατάλληλες γλώσσες και να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα. Και εδώ ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει προτείνει ένα ε, θεματολόγιο 10 σημείων ε, με πράγματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες και πρέπει να πω ότι θα μάθουμε εφαρμόζοντα τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή για να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε και την πρόσβαση στη δημόσια διαβούλευση και στη συνεισφορά πληροφοριών από όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά την αντικατάσταση, ναι, στην ε, προαρουσίασή μου προσπάθησα να τηρήσω τα πέντε λεπτά, έφτασα στα 8, πολύ εύκολα θα μπορούσα να μιλάω για 3 ώρες και η αντικατάσταση είναι βασικού και στόχη και της καινοτομίας ε, ε, και ε, της ε, επιστήμης. Η αντικατάσταση χρειάζεται προβλεψιμότητα και γνώση και αν υπάρχει προβλεψιμότητα και γνώση μπορούμε να έχουμε στοχευμένη αντικατάσταση. Συμφωνώ απόλυτα όμως ότι η αντικατάσταση είναι πάρα πολύ σημαντικός μηχανισμός στην νομοθεσία για τα χημικά για να προωθήσει την καινοτομία και επομένω να προωθήσει και την ασφάλεια. Τώρα, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τον εντοπισμό των, των ενδοκρινικών διαταρακτών και να τους απαγορεύσουμε. Η απαγόρευση είναι δική σας δουλειά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου επίσης, όχι δική μου. Και επίσης η επιτάχυνση του εντοπισμού, εδώ μπορώ να δω τρεις πτυχές οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν εμά τον Οργανισμό Χημικών Ουσιών. Ο ένα είναι να αυξήσουμε την συνέπεια και τη σχέση μεταξύ νομοθεσιών. Δεν το ε, χρειάζομαι για την νομοθεσία που εφαρμόζουμε στον δικό μα τον οργανισμό ή στην ΕΦΣΑ, γιατί υπάρχει πολύ στενή συνεργασία, αλλά θα επιταχύνει πολύ τη δουλειά μας να υπάρχουν καλύτερες συνδέσει και συνέπεια μεταξύ ημών και όλων των υπόλοιπων νομοθετικών ε, πράξεων. Ε, διαπιστώνεται για παράδειγμα ότι μια ουσία είναι ενδυνοκρινικό διαπαράκτης κάπου, είναι ενδυνοκρινικό διαταράκτης παντού. Επομένως αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Ε, ένα άλλο στοιχείο είναι ομαδοποίηση. Έτσι εμείς, όπως σας είπα, κάναμε αναδιάταξη στην υπηρεσία μας. Ε, θεωρούμε ότι η ομαδοποίηση είναι καθημερινή μας δουλειά. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά ένα μεμονωμένο χημικό στοιχείο. Και φυσικά υπάρχει... Ε, σαφής διάκριση μεταξύ του πώς μια χημική ουσία είναι διαρθρωμένη, τι ε, κοινά στοιχεία υπάρχουν μεταξύ ομάδας και τι ε, χρήσεις προβλέπονται για κάποια χημική ουσία. Ε, τα εξετάζουμε όλα αυτά και θεωρούμε ότι είναι πολύ ε, σημαντική δυνατότητα να επιταχύνουμε την ε, διαπίστωση του κατά πόσο ομοιοσία είναι ενδοκρινικός διαταράκτη. Τέλο, έχουμε τι δοκιμέ. Αν δείτε τι πληροφορίε που έχουμε και τον αριθμό των χημικών ισιών για τι οποίε χρειαζόμαστε πληροφορίε, είναι προφανέ ότι χρειαζόμαστε περισσότερε δοκιμέ και για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι ενδοκρινικοί διαταράκτε, χρειαζόμαστε περισσότερε δοκιμέ σε ζώα. Αλλά βεβαίω θα πρέπει να γίνονται δοκιμέ μόνο όταν είναι απαραίτητο για να λαμβάνουμε τη βάση για τις πληροφορίε. Αυτή είναι μια δραστηριότητα όμως την οποία λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και την οποία έχουμε επιταχύνει ουσιαστικά για τον έλεγχο συμμόρφωσης αλλά και για την αξιολόγηση των ουσιών, ε, τμήματα του REACH για να γίνονται απαραίτητες δοκιμές για να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερες ουσίες ως ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες ή να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες που είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό διότι τότε γνωρίζουμε ότι η ουσία δεν έχει τέτοια επίδραση. Τώρα, το εφέ κοκτέιλ, για να προσθέσω στα όσα είπε ο Μπέρναρτ, υπάρχουν δύο γενικοί τύποι εφέ κοκτέιλ. Υπάρχει ένα το οποίο γίνεται ε, χωρίς πρόθεση και υπάρχει και η σκόπιμη ε, διαδικασία εφέ κοκτέιλ και νομίζω ότι εσείς αναφέρεστε σε αυτό το οποίο γίνεται χωρίς πρόθεση. Η χημική νομοθεσία έχει ένα ιδιαίτερα εύρωστο πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι από τα σκόπιμα κοκτέιλ, αυτά τα οποία αποκαλούμε μείγματα, ελέγχονται καταλήλως. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά διότι θα πρέπει να γίνει ομαλή και αποτελεσματική διαπαφή μεταξύ, για παράδειγμα, της ε, ε, επισήμανσης και της ε, ταξινόμησης και την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο της εργασίας που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Επίσης, σε συνέχεια των όσων είπε ο Μπέρνερ, το βασικό είναι να δούμε ποια είναι ε, τα, ε, τα εφέ κοκτέιλ τα οποία δεν έχουν γίνει από πρόθεση. Και εδώ νομίζω ότι αυτό το οποίο ε, συμβάλλει πολύ σε αυτά τα εκούσια εφέ κοκτέιλ είναι το να συλλέξουμε τα ε, δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά επίσης ε, να καθοδηγήσουμε και προς νέα στοιχεία παρακολούθησης και για την παρακολούθηση ανθρώπων, αλλά και παρακολούθηση στο περιβάλλον και στα άγρια είδη, κάτι το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά. Σαφώς λοιπόν η διαδικασία της ομαδοποίησης ε, θα βοηθήσει. Έχουμε, ε, όπως και οι συνάδελφοι στην ΕΦΣΑ, ε, Έχουμε κάνει κάποια δουλειά για ε, εκούσια έκθεση σε εφέ κοκτέιλ, όπως και οι συνάδελφοι στην ΕΦΣΑ. Και ε, υπάρχει λοιπόν ε, μια βάση ε, και το νομικό πλαίσιο στην νομοθεσία για τα χημικά μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά μας ενδιαφέρει και η βάση, η οποία όπως εξήγησε και ο Μπέρναρτ, είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως. Τέλος, να μιλήσω για τα τέλη και τους πόρους. Και πάλι η, τα τέλη δεν είναι δική μας δουλειά. Το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση μόνο από τα τέλη ή όχι είναι πολιτική απόφαση, διότι εκεί σταθμίζουμε πώς εσείς θέλετε να ε, εφαρμόσετε την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει και το πώς επιβαρύνει ένα τέτοιο τέλος στη βιομηχανία. Αυτό λοιπόν δεν είναι δικό μας ε, πεδίο. Ε, είναι ε, θέμα πολιτικής. Εμείς ε, δυσκολευόμαστε να έχουμε εισοδήματα από τα τέλη, αλλά αυτό είναι ε, μια σημαντική πτυχή που αφορά τον προπολογισμό. Μπορώ πολύ ευχαρίστω να το εξηγήσω, αλλά ίσω όχι τώρα. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν θεωρούμε σε καμία περίπτωση ότι είμαστε στο τσεπάκι τη βιομηχανία γιατί μα πληρώνουν τέλη. Εμεί θεωρούμε από πλευρά μα ότι είναι η δική μα η επιλογή ε, να αποφασίζεται πώ θα καταβάλλονται τα τέλη ή όχι προ την ε, υπηρεσία χημικών ουσιών. Τώρα, όσον αφορά το σπόρου, το ερώτημα είναι τι θέλετε να κάνουμε και θα σα πω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Αν, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι θέλετε να εφαρμόσουμε πλήρω τι δράσει στην αναθεώρηση του ΡΙΤΣ, να τα επιταχύνουμε και να τελειώσουν μέχρι το 2027, να επιταχύνουμε τη δουλειά για τι αδειοδοτήσει, του περιορισμού, ε, τα βιοκτώνα και τη δουλειά μας για την ομαδοποίηση, που είναι ουσιαστικά τα πολιτικά μηνύματα που λαμβάνουμε, τότε χρειαζόμαστε σταθερούς πόρους. Μπορώ να επιταχύνω με σταθερούς πόρους και με προβλέψιμους πόρους. Το καθεστώ του περιβότου δελτίου 32 που ήταν το βασικό στοιχείο για τι υπηρεσίε, δεν μα ε, παρέχει μια τέτοια βάση αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αυτή την πρόταση πριν από τι νέε πολιτικέ προτεραιότητε. Αν δούμε όμω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση των υπηρεσιών και των οργανισμών και τη δική μου τη υπηρεσία. δεν έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο βάση του οποίου μπορούμε να εφαρμόσουμε τι ε, πολιτικέ, ε, όπω βλέπετε για παράδειγμα και στον έλεγχο στο fitness Τη της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και δεν μπορούμε να συμβάλλουμε και να σε οποιαδήποτε προσαρμογή που θα προέλθει από το fitness check όλες τις νομοθεσίες για τα χημικά πέραν του REACH. Για να κάνουμε λοιπόν αυτά που έχουμε τώρα, ε, χρειαζόμαστε σταθερούς πόρους, συνέχεια αυτών που έχουμε τώρα, προφανώς ε, θα πρέπει να γίνει και προσαρμογή προς τον πληθωρισμό και αν θέλετε να κάνουμε περισσότερα, τότε θα χρειαστούμε ε, και θέλουμε περισσότερους πόρους πέραν αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, και κάτι την ε, διάρκεια του κοκτέιλ, του πραγματικού κοκτέιλ, έτσι με ποτά, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε περαιτέρω αυτά τα ζητήματα. Περνάμε τώρα ε, στο δεύτερο τμήμα εδώ τη ε, συζήτηση με του οργανισμού ε, και τώρα έχουμε τον Οργανισμό Φαρμάκων, τον EMA και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, το ECDC. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Οργανισμό Φαρμάκων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ εδώ τα αξιότιμα μέλη που μα δίνουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις σκέψεις μας και να παρουσιάσουμε τον τρόπο που λειτουργεί. Λειτουργούν αυτοί οι πέντε οργανισμοί. Που επίπνουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν λίγο το πώς λειτουργούμε και ζητώ βέβαια συγγνώμη εκ των προτέρων από εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το τι κάνουμε και μας παρακολουθούν εδώ και χρόνια στις εργασίες μας. Αλλά νομίζω πως θα είναι χρήσιμο το να αναφέρουμε έτσι κάποια βασικά στοιχεία ως προς το τι ακριβώς θα κάνουμε. Επί της αρχής λοιπόν παρέχουμε μια επιστημονική αξιολόγηση όλων των καινοτόμων φαρμακευτικών συσκευασμάτων για έγκριση σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Δηλαδή, Ουσιαστικά 500 εκατομμύρια πολίτες μέσω μία αίτηση μπορούν να υποβληθούν σε μια αξιολόγηση και να λάβουν μια άδεια η οποία ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζουμε λοιπόν τα ίδια πρότυπα, έχουμε στην ίδια χρονική στιγμή, όπου αυτό χρειάζεται δηλαδή, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Τι περιλαμβάνεται εδώ στο, στην εντολή μας. Κυρίως καινοτόμα φάρμακα, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη μετώπιση του καρκίνου, ε, της μόλυνσης με τον ε, ιό ανθρώπινης ε, το, τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, αλλά και τις νέες καινοτόμες θεραπείες, για παράδειγμα σε επίπεδο γονιδίων και σε κυταρικό επίπεδο. Επίσης, προωθούμε την καινοτομία μέσω επιστημονικής, επιστημονικών συμβουλών, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να παραχθούν τα απαραίτητα στοιχεία, επιστημονικά στοιχεία, τα οποία θα μας επιτρέψουν να αντιοδοτούμε νέα φάρμακα. Και αυτό θα επιτρέψει βέβαια την διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, χωρούς, σε ασθενείς δηλαδή, χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι που θα συνοδεύουν αυτές τις δοκιμές. Ένας ακόμα ε, σημαντικός πυλώνας βέβαια της δραστηριότητάς μας εδώ είναι η ασφάλεια. Δηλαδή ε, παρακολουθούμε από κοντά και στενά ε, περισσότερα από μισό εκατομμύριο φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά της Ένωσης. Να σας πω όμως τι δεν κάνουμε, την συγκαταλέγεται στη δική μα εντολή. Δεν δίνουμε εγκρίσει ό,τι αφορά τι κλινικέ δοκιμέ, γιατί αυτό το εγκρίνουν τα κράτη-μέλη, πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Και επίση δεν λαμβάνουμε καμία απόφαση σε ό,τι αφορά είτε την τιμή, είτε τι αποζημιώσει για την ε, πλήρωμε τον, ε, τις ε, τιμής των φαρμάκων. Και αυτά τα ζητήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατομέλων. μελών. Τι, πώς όμως, ποια είναι η σύνθεσή μας. Είμαστε μια σχετικά, ένα σχετικά μικρός οργανισμός με γύρω 500 άτομα ως προσωπικό αν το συγκρίνουμε αυτό με τους 8.000 για παράδειγμα του Οργανισμού Φαρμάκων του Ηνωμένων Πολιτειών και τις 5.000 της Ιαπωνίας θα διαπιστώσετε ότι είμαστε μια σχετική, σχετικά μικρή υπηρεσία, ένα σχετικά μικρός οργανισμός. Ε, και πώς ε, επιτυχάνουμε να έχουμε τόσο μικρό αριθμό προσωπικό. Το κάνουμε επειδή έχουμε ένα δίκτυο και ένα κοινό πουλ από 55 εθνικές αρχές και υγειονομικές και εκτινεατρικές ε, μέσω των οποίων έχουμε ήδη προεγκεκριμένους πάνω από 4.000 εμπειρογνώμονες από την δική τους ε, πλευρά ε, οι οποίοι έχουν δηλαδή προελεγχθεί και για περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων και την εμπειρογνώμοσύνη του. Ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί κανένα κράτο μέλο δεν έχει τη δυνατότητα να διατηρεί για παράδειγμα 4.000 εμπειρογνώμονε, ε, οι οποίοι ακριβώ ε, θα ανανεώνονται συνεχώ και θα λαμβάνουν περισσότερες γνώσει. Έχουμε από εκεί λοιπόν και μετά πέραν από αυτού του εμπειρογνώμονε, 7 επιστημονικέ επιτροπέ και από εκεί και μετά βέβαια μα υποστηρίζουν και επιστημονικέ συμβουλευτικέ ομάδε και ομάδε εργασία εμπειρογνώμονων. Τώρα, επιτρέψτε μου να σα εστιάσω λίγο στι συγκεκριμένε δραστηριότητε που αναλαμβάνουμε σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη ασφάλεια. Πέρυσι λάβαμε 2 εκατομμύρια περιπτώσεις ή αναφορές παρενεργειών. Και με βάση τα όσα λάβαμε, καταφέραμε να εστιάσουμε στο τι ακριβώς τελικά συμβαίνει σε επίπεδο παρενεργειών ε, και τι όχι και με βάση τα όσα εμ, διαπιστώνουμε αποσύρουμε κάποια φάρμακα από την αγορά ή αλλάζουμε την, ε, ε, τον τρόπο χρήση τους και τη δοσολογία ακριβώς βασιζόμενοι σε αυτή τη συνεχή παρακολούθηση. Και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τέτοια κρούσματα διαπιστώνουμε ότι δεν σχετίζονται τελικά με τη χρήση του συγκεκριμένου φαρμάκου. Και αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό, αποτελεί ουσιαστικά τον ακρογωνίο λίθα, αν θέλετε, για την ασφάλεια, αλλά δεν υπάρχει από μόνο. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε και άλλες προσπάθειες. Γιατί βλέπουμε τώρα να υπάρχει μια ε, νέα γενιά φαρμάκων, κυταρικών λοιπόν και γονιδιακών, ε, που μπορούν να μεταλλάξουν, αν θέλετε, να αλλάξουν οριστικά τις ιδιότητες του σώματος του ασθενούς, ο οποίος θα λαμβάνει. Για γι' αυτό λοιπόν ακριβώς θα πρέπει ήδη στο επίπεδο ε, του σχεδιασμού του φαρμάκου θα πρέπει να προβλέπεται το ζήτημα της ασφάλειας εφόρου ζωής για τον ασθενή. Οπότε εδώ αλλάζει εντελώς η σκέψη, η συλλογιστική την οποία ακολουθούμε και θα πρέπει βέβαια να παρακολουθούμε και τις ε, εξελίξεις τις τεχνολογικές. Εδώ αναφέρομαι ειδικότερα στη τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνεχής παρακολούθηση και ε, ε, εμπειρία πραγματική σε ό,τι αφορά την, την, τις επιδόσεις του φαρμάκου, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση γρήγορα να αντιδρούμε και να μετατρέπουμε αναλόγως το, κανονιστικό πλαίσιο. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό πάντοτε να λαμβάνεται ε, υπόψη και η τοποθέτηση των πολιτών και του, του, του ΕΣΑ δηλαδή για την ασφάλεια των τροφίμων. Επίσης προσπαθούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για το μέλλον. Όπως ε, μπορείτε να φανταστείτε είναι καταρχήν και σε επίπεδο νομοθετικό έχουμε τέσσερις κανονισμούς. Καταρχήν το κανονισμό σε ό,τι αφορά τις κλινικές δοκιμές γιατί θα υπάρξουν και κλινικέ δίκαιε οι οποίε θα τρέχουν, ε, θέλουμε να τρέχουν παράλληλα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα ίδια πρότυπα και με έναν πιο βελτιστοποιημένο τρόπο και με την παροχή περισσότερων εγγυήσεων προ τον ασθενή. Και όλα αυτά με πιο αποδοτικό, αποτελεσματικό τρόπο. Μετά έχουμε τον, την ε, νέα νομοθεσία, τον κανονισμό σε ό,τι αφορά την, τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε 56 λοιπόν διαφορετικέ βάσει δεδομένων οι οποίε περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα ασθενών. Πράγμα βέβαια το, το οποίο θα αποτελέσει μια μεγάλη πρόκληση για μας προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και θα υπάρξει και βέβαια κάποιο ζήτημα σε ό,τι αφορά την δευτερογενή, αν θέλετε, χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων. Και θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις έτσι ώστε να βρούμε μια σωστή λύση με τις ε, σχετικέ αρχές. Μετά, ο κανονισμός σε ό,τι αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα γιατί ε, όλο και περισσότερο αναφερόμαστε σε διαδικασίες και σε όχι στα φάρμακα αυτά καθεαυτά Δηλαδή ε, στο μέλλον η διαφορά ανάμεσα σε ένα τεχνολογικό προϊόν και σε ένα φάρμακο θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα περιπτώσεις εχείρησης όπου έχουμε μοσχεύματα σε ε, ύπαρη ή οτιδήποτε άλλο με τη χρήση νανοτεχνολογίας, ε, οι συσκευές οι οποίες ακριβώς εμφυτεύονται μέσα στο ανθρώπινο σώμα και ούτω καθεξής αποτελούν παραδείγματα για αυτήν την, την, το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφές πλέον όριο ανάμεσα σε αυτά τα προϊόντα και τα φάρμακα. Αυτή λοιπόν η, η αλλαγή που λαμβάνει η χώρα στην τεχνολογία ε, θα αρχίσει να απαιτεί και μια αντίστοιχη αλλαγή στην νομοθεσία και κατά συνέπεια θα πρέπει ήδη από τώρα να προετοιμαζόμαστε. Και βέβαια ταυτόχρονα ανακύπτει εδώ και το, το, το ζήτημα της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης. Επίσης θα πρέπει να ε, προετοιμαστούμε σε ό,τι αφορά δύο κυρίως ζητήματα. Καταρχήν η ψηφιακή ε, μεταμόρφωσε. Γιατί το 2016 ήμασταν ήδη παροχημένοι αν θέλετε, ενώ τώρα πια ε, θεωρούμαστε δύο αρχαίοι αν θέλετε ε, ως προς την ε, προσέγγιση που ακολουθούμε. Και αυτό επειδή δεν είχαμε θέσει τις σωστές προτεραιότητες. Και Ε, δεν θα πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να επανέλθουμε στα επίπεδα που βρισκόμαστε στο 2016. Τώρα, τι κάνουμε στο πλαίσιο της ε, πολύ συγκεκριμένης εντολής ε, που έχουμε. Ξέρουμε τι κάνει το μοντέλο με βάση το οποίο λειτουργούμε και τι επιτυγχάνει, αλλά ε, μας ε, ενοχλεί το γεγονός ότι ε, εγκρίνουμε πολλά φάρμακα, αλλά όλο είναι και περισσότερο, λιγότεροι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε αυτά γιατί η, τα ζητήματα τιμής είναι εκείνα που δημιουργούν ακριβώς όλο ένα και μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στην έγκριση αφενός και την πραγματική πρόσβαση των ασθενών σε ένα φάρμακα αφετέρου. Άρα λοιπόν εδώ κάνουμε, έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία ώστε να δούμε ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος κατανομής των διαθέσιμων ε, πόρων και πώς μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Όπως σας είπα, ε, προετοιμαζόμαστε όλο και καλύτερα σε ό,τι αφορά αυτά τα νέα φάρμακα ή θεραπείες καλύτερα να τα πούμε έτσι και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις ελλείψεις σε ό,τι αφορά τα φάρμακα δηλαδή που πλήττουν πολλές χώρες της Ένωσης αλλά και εκτός αυτής για πολλούς λόγους και μπορώ να επεκταθώ σε αυτό και περαιτέρω. Και επίσης ε, υπάρχουν όλο ένα και περισσότερα προβλήματα που προκύπτουν σε ό,τι αφορά την αλυσίδα του εφοδιασμού. Δηλαδή, ε, το 85% της αλυσίδας ε, αγωγής αυτών των φαρμάκων έχει τουλάχιστον ένα σκέλος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πράγμα το οποίο δημιουργεί όλα τα θετικά ζητήματα λασιμότητας και παρακολούθηση της ποιότητας των ελόγων φαρμάκων. Και επίσης θέλουμε και εμείς από την πλευρά μας να συμβάλλουμε στην επίλυση του ζήτηματο τη μικροβιακή αντοχής αλλά και τη απροθυμίας ορισμένων ε, για τους εμβολια... απέναντι στου εμβολιασμού. Αυτά από την δική μου πλευρά θα σταματήσω εδώ και με τα χαρά να ακούσω ερωτήματα. Ευχαριστούμε για το ECDC τώρα, η κυρία Μον. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αξιότιμοι προβουλευτές, το 2003 ξεκινήσαμε όταν ε, νέες ασθένειες ε, με ανησυχητική ταχύτητα επεκτάθηκαν στην Ευρώπη. Και τότε φάνηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται οργανισμό που να συλλέγει τα στοιχεία για τις αναδιόμενες αυτές ασθένειες σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και να μπορεί να τα αξιολογεί. Έτσι εγκρίθηκε νομοθεσία πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με το τι ήθιστε και το 2005 έτσι δημιουργήθηκε και άρχισε να λειτουργεί ο... το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Εκτός από το Λουξεμβούργο, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη εκπροσωπούνται. Οπότε σιγά σιγά στο κέντρο μας ενσωματώθηκαν όλοι. 62% του προσωπικού μας είναι γυναίκες και 38% είναι άντρες. Οπότε βλέπετε το νέο μας κτίριο εδώ, ε, όπου εγκατασταθήκαμε εκεί τον Απρίλιο που μας πέρασε. Λοιπόν, η αποστολή μας και ο ρόλος μας είναι να εντοπίζουμε, να αξιολογούμε και να επικοινωνούμε τρέχουσες και αναδιόμενες απειλές για την ανθρώπινη υγεία από μολυσματικές ασθένειες. Βλέπετε εδώ λοιπόν ποια είναι τα κύρια καθήκοντά μας και τις διάφορες ομάδες ασθενειών πάνω στις οποίες εργαζόμαστε και τα τελευταία χρόνια είχαμε και ένα νέο κατάλογο ασθενειών που παρακολουθούμε και είναι τώρα 57. Οι κύριες προτεραιότητές μας είναι η μικροβιακή αντοχή και εμείς πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε περισσότερα αποτελέσματα ακόμα όταν έχουμε ιδιαίτερε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα είχαμε την Ιλαρά. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες μέλη εργάζονται προκειμένου να ε, επιτευχθούν οι στόχοι μας και να καταπολεμιστούν ασθένειες όπως το AIDS και η πατήτιδα. Συνεργαζόμαστε με τις χώρες μέλη, με δίκτυα και προσφέρουμε επιδημιολογική ανάλυση τα στοιχεία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να τα βρει. Ε, δίνουμε επίσης κατευθυντήριες ε, γραμμές όσον αφορά την επικινδυνότητα. Τώρα, αν πάτε στην ιστοσελίδα μας και στο κέντρο ε, για επίγουσα ανάγκη, βλέπετε ότι οι συνάδελφοι συναντιόνται κάθε μέρα και σε καθημερινή βάση ελέγχουμε τις εξελίξεις και αξιολογούμε τις απειλές. Και αυτό το κάνουμε κοιτώντα τη συνολική εικόνα. Γιατί οτιδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη σε 24 με 48 ώρες. Τίποτα δηλαδή δεν βρίσκεται πολύ μακριά από μας. Συλλέγουμε λοιπόν και αναλύουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες. Τώρα, σε, αυτό, σε αυτή τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, καθημερινά λαμβάνονται αποφάσεις. Κατά πόσο θα παρακολουθήσουμε ε, κάποια υπόθεση, κάτι μπορούμε να το αφήσουμε απ' έξω, για κάτι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες ή για κάτι χρειάζεται πραγματικά αξιολόγηση κινδύνου. Τι κίνδυνος δηλαδή μπορεί να ελοχεύει στην Ευρώπη ή σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης ή ε, τι μπορεί να μπει μέσα στην Ευρώπη από κάποιον ο οποίος θα έρθει από κάποια περιοχή. Η αξιολόγηση αυτή κινδύνου γίνεται μέσα σε λίγες μέρες με πυρογνώμονες και από την εκάστοτε χώρα και η αξιολόγηση κινδύνου περιλαμβάνει και κάποιες δυνατότητες αντιμετώπισης. Το καλύτερο λοιπόν ε, που κάνουμε είναι αυτή η αξιολόγηση κινδύνου και αυτό είναι που εκτιμάει ο κόσμος πάρα πολύ από το έργο μας. Μερικοί μάλιστα που κάνουν την αξιολόγηση κινδύνου από μόνοι τους έχουν σταματήσει να το κάνουν γιατί βασίζονται στις δικές μας αξιολογήσεις κινδύνου. Φυσικά και υπάρχει και συντονισμός και στήριξη σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές ε, επίπεδο. Εμείς στηρίζουμε βέβαια όταν διασυνοριακά προκύπτει κάποιος κίνδυνος, αλλά και σε εθνικό επίπεδο επίσης. Ένας από τους εμπειρογνώμονές μας βρίσκεται τώρα στο Κονγκό. για την αντιμετώπιση του έμπολα. Έχουμε φυσικά και εταίρους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρε μέλη, οι άλλε υπηρεσίε και οργανισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και έχουμε επίση και εταίρου εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κυρίω η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, βέβαια, με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με το Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Γραφείο τους. Επίσης με τις χώρες διεύρυνσης και γειτονίας και υπάρχει τώρα μια μεγάλη διάσκεψη στη Γεωργία με τις χώρες διεύρυνσης και γειτονίας, όπου συζητάμε τα θέματα υγείας και την μικροβιακή αντοχή συζητάμε συγκεκριμένα στην Γεωργία τώρα και προσπαθούμε να δούμε πώς θα ενισχύσουμε το έργο που γίνεται για την μικροβιακή αντοχή, την αντοχή δηλαδή σε αντιμικροβιακά φάρμακα ε, στις χώρες αυτές. Συνεργαζόμαστε φυσικά και με άλλες χώρες ανά τον κόσμο και προσπαθούμε να συγκρίνουμε και την κατάσταση όσον αφορά το μέγεθος και τον προπολογισμό σε εμά και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μπορώ να σας δώσω για να μην νομίζετε ότι εδώ καθόμαστε ένας δίπλα στον άλλον, ωραία και καλά και δεν κάνουμε τίποτα. Όχι, συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Έχουμε μια έκθεση που εκπονούμε με την Υπηρεσία Φαρμάκων και με την ΕΦΣΑ για την κατανάλωση ε, των ε, φαρμάκων ε, και την μικροβιακή αντοχή. Και πόσο γνωρίζω, είναι ο μόνος ε, τομέας ε, στον ε, κόσμο που καλύπτει τόσο μεγάλη γεωγραφική επιφάνεια και πληθυσμό με ολοκληρωμένη ανάλυση. Έγινε το 2015 και 2017 και τώρα ετοιμαζόμαστε για του χρόνου να έχουμε την νέα εκδοχή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους αρμόδιους ε, επαφής της ΕΜΒΗ για το κάθε οργανισμό. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπουσέο για τον Οργανισμό Φαρμάκων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Καμφάν. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και συγχαρητήρια στους πέντε οργανισμούς και υπηρεσίες για την επιτεύγματά σας. Είναι τιμή μου να είμαι το σημείο επαφή ε, για τον Οργανισμό Φαρμάκων, που είναι μία από τις επιτυχημένε ιστορίες στον τομέα της υγείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δραστηριότητες στην ανθρώπινη υγεία και στον κτηνιατρικό τομέα ε, δίνουν τη δυνατότητα για πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα που σώζουν ζωές ε, στους Ευρωπαίους πολίτες ε, νωρίτερα από ό,τι πριν, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και ψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Δύο συγκεκριμένε ερωτήσεις, δύο συγκεκριμένα θέματα, τα οποία θα ήθελα να απευθύνω στον κύριο καθηγητή, τον Γκουίντο Ράζη, όσον αφορά τι μελλοντικέ προκλήσει. Μία από τις προκλήσεις είναι η μετεγκατάσταση στο Άμστερνταμ. Αν δεν κάνω λάθο, ετοιμάζεστε να ε, μετακομίσατε στο τελικό κτίριο αρχές του ερχόμενου έτους. Αλλά αν κατάλαβα καλά, στη διαδικασία της μετακόμισης από το Ηνωμένο Βασίλειο, σημαντικός αριθμός ε, του δυναμικού του οργανισμού αποχώρησε. Φοβάμαι ότι ο οργανισμός ε, δεν θα έχει απαραίτητους ανθρωπίνους πόρους προκειμένου να διεξάγει όλα τα καθήκοντά του και λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και θα το ανατεθούν μετά από την νομοθεσία που ε, ψηφίστηκε τα τελευταία χρόνια. Πώς έχει η κατάσταση και τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να σας υποστηρίξουμε για να επιλύσετε αυτή την κατάσταση. Και το δεύτερο αφορά το GDPR. Προφανώς και η νέα νομοθεσία είχε σημαντικό αντίκτυπο για την καθημερινή μας ζωή. Χρειαζόμαστε καλή προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με τη νέα νομοθεσία η προστασία αυτή ενισχύθηκε, αλλά συζητώντας ε, με πολλούς ε, εκπροσώπους πανεπιστημίων, πολλούς εκπροσώπους ε, Τη ερευνητικό κοινότητα ε, τη Ευρώπη και τη χώρα μου, τη Ρουμανία, ε, αντιλαμβάνομαι ότι η νέα νομοθεσία μπορεί να έχει και αρνητικό αντίκτυπο για την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων και για την έρευνα για την υγεία εν γέννη. Μπορείτε να μας πείτε σας παρακαλώ ποιες είναι οι συνέπειες του GDPR για τη δική σας τη δουλειά στον EMA και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα μετά από την ε, εφαρμογή πλέον της νομοθεσίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες. Ευχαριστώ και για το ECDC η Γιάννα Κοσμίσκα από το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα ε, του εκπροσώπους του ECDC για τη χθεσινή συνεδρίαση. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πραγματικά ε, πλήρη ε, περιεχομένου. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό οργανισμό, ιδιαίτερος τώρα που συζητούμε και πάλι τον έμπολα, για παράδειγμα. Και αυτό είναι και μία από τις ερωτήσεις μου. Πώς ε, μπόρεσε το ECDC να παρακολουθήσει την επιδημία που είχαμε ε, στην Ιταλία. Ε, εχθές ε, συζητήθηκε και το ψήφισμα για τη διευκόλυνση της ε, ε, παροχής ε, ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης. Και βάσει του ψηφίσματος πρέπει να γίνεται καλύτερη προαγωγή της υγείας και πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε περίπτωση πανδημίας. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν εχθές και ακούσαμε πόσο σημαντική ήταν η δραστηριότητα του οργανισμού ε, στη διάρκεια της παρουσίασης. Έχω μία ερώτηση. Πώς βλέπει ο οργανισμός ε, μια στενότερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τομείς. Αν ναι, ε, ποιοι είναι αυτοί οι τομείς ε, και πού θεωρείτε ότι θα μπορούμε να έχουμε στενότερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο και στους υπολείπους ο κύριος Λουένα. Ξεκινάμε μαζί σας. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο. Είναι σαφέ από αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί ότι ο προπολογισμό ε, των οργανισμών και των υπηρεσιών θα πρέπει να αναθεωρηθεί και μάλιστα σύντομα. Διότι είναι προφανέ ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα ή τουλάχιστον μια στρέβλωση. Κάποιοι από εσά είπαν ότι αυτό βέβαια επαφείται στου πολιτικού. Ε, ναι, Στου ευρωβουλευτέ και στα μέλη του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τουλάχιστον από την ομάδα μα θα είναι χαρά να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μια συγκεκριμένη ερώτηση τώρα ε, στον κύριο Ράτσι για τον Οργανισμό Φαρμάκων, για τη συμμετοχή του κλάδου σε αυτόν τον οργανισμό είναι, προσοχή εδώ, το 90%. Η ερώτησή μου είναι, έχει αυτό σχέση αιτίου αποτελέσματος ε, ε και δείχνει ότι δεν υπάρχουν πραγματικά καινοτόμα φάρμακα διότι η σύνθεση και ο προϋπολογισμός ε, του οργανισμού είναι κατά 90% από τον κλάδο και μόνο 10% από το δημόσιο προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ, ο κύριος Πόζακ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Και εγώ έχω μια ερώτηση για τον προπολογισμό. Με κάλυψε βέβαια ο προλαλή σα. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί και οι υπηρεσίε κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και το εκτιμώ. Οι ανάγκε τώρα προ τον προπολογισμό μπορεί και να είναι απεριόριστε σε κάποιες περιπτώσεις. Επομένως, έχουμε δικαίωμα να ελέγχουμε τον προπολογισμό και να γίνει το κατάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχος, ώστε οι δαπάνες τους να είναι βιώσιμες. Θέλω να, να ρωτήσω για την καταπολέμηση του καρκίνου. Η εκλεγήσα πρόεδρος Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι αποτελεί προτεραιότητα το θέμα του καρκίνου και για κάποιους είναι πανευρωπαϊκό το θέμα αυτό. Και θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και οι υπηρεσίες θα πρέπει να βοηθούν προ αυτή την κατεύθυνση. Είστε λοιπόν διατεθειμένοι να ασχοληθείτε με αυτή την προτεραιότητα βάση και του προπολογισμού που διαθέτετε και μπορείτε να καταπαλωμήσετε καλύτερα τον καρκίνο γιατί αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα θητεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ευχαριστώ. Η κυρία Κονιέτσινα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συναδελφοί, τα τελευταία πέντε χρόνια ήμουνα το σημείο επαφή για το ECDC και θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στη συνάδελφο που έχει αναλάβει το θέμα και πραγματικά φροντίστε τον ECDC γιατί είναι εξαιρετικός οργανισμός για να του φερθείτε καλά. Είναι η πιο μικρή υπηρεσία που έχουμε, αλλά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και με πολύ λίγα χρήματα. Και συμφωνούμε εδώ ότι δεν είναι μόνο ο οργανισμός φαρμάκων αυτός ο οποίος δουλεύει, αλλά και ο ECDC μας προστατεύει από μολυσματικές ασθένειες, τις οποίες ευτυχώς ακούμε μόνο στην τηλεόραση, αλλά υπάρχουν. Και μπορεί να δράσει άμεσα, έχει τεράστια εμπειρογνωμοσύνη σε όλη την Ευρώπη και πολύ συχνά το λησμονούμε. Από την άλλη, θεωρώ ότι δεν είναι μόνο καρκίνος, αλλά υπάρχουν και θέματα όπως ε, οι εμβολιασμοί, είναι θέμα το οποίο αφαιρά άμεσα τον ECDC. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πράγματα για τον εμβολιασμό και τη μικροβιακή εντοχή, πώ να αντιμετωπίσουν τα θέματα εμβολιασμού σε διάφορε χώρε και τι απειλή ε, υπάρχει για του πολίτε μα στην Ευρώπη. Ελπίζω λοιπόν να δοθεί προτεραιότητα στα θέματα αυτά, στους οργανισμού αυτά, για τους, γιατί του αξίζει. Υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων η οποία μας προσφέρει υλικό, μας δίνει πληροφορίες, μας συνεργάζονται μαζί μας και πιστεύω ότι δεν είμαστε πάντα σε θέση να δεχτούμε ό,τι προσφέρουν. Χαίρομαι λοιπόν που τα εξετάζουμε ακόμα, προσέχουμε, αναζητούμε πληροφορίες και δεδομένα και μάλιστα σε... Ε, εκεί που υπάρχουν. Και αν ε, προσέχουμε λίγο περισσότερο τους οργανισμούς και ε, διαβάζουμε τις εκθέσεις, ε, θα κερδίσουμε χρόνο και ενέργεια. Ευχαριστώ και να πω και πάλι στο ECDC ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και παρά το γεγονό ότι δεν είμαι πια το άτομο επαφή μαζί του, θα αποτελούν και πάντα θα αποτελούν προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλο κανεί. Όχι. Νομίζω λοιπόν τώρα ότι μπορούμε να περάσουμε στι απαντήσει προ τι ερωτήσει. Ξεκινάμε με τον ECDC. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Για το πώς παρακολουθούμε επιδημίες. Έχουμε διάφορα εργαλεία για αυτό το σκοπό. Οι επιθυμίες αυτές συνήθως ε, τη χάνουν παρακολούθησης από άμεσες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη, διότι Γιατί ορισμένε φορέ ε, τα στοιχεία παρακολούθηση καθυστερούν. Υπάρχουν όμω συστήματα τα οποία μα επιτρέπουν να διαπιστώσουμε που έχουμε πληροφορίε και έχουμε και δίκτυα ε, τα οποία μα δίνουν άμεσα πληροφορίε. Υπάρχει στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη σε όλους τους τομείς της εντολής μας. Όπως σας είπα, μέσω των δικτύων υπάρχουν ε, εθνικά σημεία εστίασης για συγκεκριμένες ε, νόσους ή ομάδες ε, νόσων και ασθενειών και υπάρχει πάρα πολύ στενή συνεργασία μεταξύ μας. Θεωρούμε ότι υπάρχει και κάτι θετικό στις επισκέψεις σε κάθε χώρα, διότι αφενός είναι πάρα πολύ σημαντικό από πλευράς πόρων και για το κράτος και για μας, αλλά μπορούμε να μάθουμε τα καλύτερα πράγματα για μια χώρα, για ένα συγκεκριμένο τομέα, ώστε να προσφέρουμε και εναλλακτικέ λύσεις για δράσεις οι οποίες στοχεύουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι όπου επιθυμούμε να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία, να έρθουν σε επαφή μαζί μας τα κράτη-μέλη και να έχουμε τέτοιες επαφές και αν είχαμε περισσότερους πόρους ε, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε για να έχουμε πιο στοχευμένη στήριξη για τα κράτη-μέλη. Για τον καρκίνο, όπως ανέφερα, η εντολή μας αφορά μολυσματικές ασθένειες. Υπάρχουν ε, καρκίνοι οι οποίοι προκαλούνται από μολυσματικές ασθένειες, όπως για παράδειγμα από μόλυνση από υπατήτιδα, ή από τον HPV, ε, έχουμε καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ε, εδώ υπάρχουν κάποια στοιχεία, αλλά δεν συλλέγονται στοιχεία για τον καρκίνο και δεν είναι τμήμα της εντολής μας. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, πρώην, ε, το πρώην άτομο επαφής, την κυρία Κονέτσια. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. EMA. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέσσερις ερωτήσεις θυμάμαι. Φόρτος εργασίας και πόρη. Και τι γίνεται με την ε, μετακόμισή μας. Να πω ότι υπάρχουν δύο πτυχές. Αυτή που είχαμε το 2016, όταν ξεκίνησε αυτή η μακρά διαδικασία της μετεγκατάστασης λόγω Brexit, είναι 120 λιγότεροι. Έφυγαν όλοι αυτοί οι προσωρινώς εργαζόμενοι, τους οποίους δεν μπορούμε να τους ξαναπροσλάβουμε λόγω διαφορετικού εργατικού δικαίου εκεί που εργαζόμαστε. Επομένως θα πρέπει να φτάσουμε στο εργατικό δικαιονομικό του 2016. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ανησυχία για μας. Μετά, μας έχουν αναθέσει τέσσερα νέα καθήκοντα και πριν από αυτό έγινε περικοπή 60 θέσεων. Ο προπολογισμό μας που κατά 95% προκύπτει από τη δική μας τη δραστηριότητα ανέβηκε κατά 38%. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες θα πληγεί σίγουρα η ποιότητα, είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο, ε, ε, επομένως η παρακολούθηση και η ποιότητα των επιστημονικών διαγνωμοδοτήσεων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα ε, στο μέτρο του δυνατοτήτων μας. Μέχρι τώρα έχουμε σεβαστεί τα χρονοδιαγράμματα, το 100% των περιπτώσεων, εκτός από κάποιες καθυστερήσεις ε, για κάποια πιστοποιητικά και κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με τη δημόσια υγεία. Το σύστημα πληροφορικής μας έχει αρχίσει να ε, είναι παλιό και φυσικά το τίμημα θα το πληρώσουμε σε 3-4 χρόνια. Θα υπάρχει πλήγμα στη διαφάνεια, υπάρχει καθυστέρηση στην πρόσβαση των εγγράφων και Βρισκόμασταν στην πρώτη γραμμή της διαφάνειας. Ήμασταν ο πρώτος οργανισμός παγκοσμίω που δημοσίευε τα στοιχεία των κλινικών δοκιμών μετά από ένα μεγάλο πόλεμο. Δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα όμως να συνεχίσουμε τη δημοσίευση. Αυτά λοιπόν καθυστερούν. Εν τω μεταξύ, οι αρχές του Καναδά και άλλες αρχές ακολουθούν το παράδειγμά μας και αυτό είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό. Πώς θα αντιμετωπίζουμε τώρα. Έχουμε δύο task force οι οποίες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη ρομποτική και την ψηφιοποίηση όσο περισσότερο γίνεται για να έχουμε κάποιους πόρους για νέες δραστηριότητες, αλλά όλα αυτά είναι μακροπρόθεσμα, αφορούν την ε, χρηστή διαχείριση και το σχεδιασμό όλα αυτά και όπως σας είπα ε, αυξήθηκε ο προπολογισμό μας με μηδενικό κόστος ε, για τις δημόσιες δαπάνες. Είναι ανοησία λοιπόν όλα αυτά, αν μου επιτρέπετε. Και αν μου επιτρέπετε επίσης, θα ήθελα να περάσω και στην άλλη ερώτηση για τα τέλη από τη βιομηχανία. Και θα επανέλθω μετά στο θέμα του GDPR. Για όσους δεν γνωρίζουν όλο το μηχανισμό, φαίνεται πολύ περίεργο να εξαρτάται κάποιος ε, από τα τέλη, από το κλάδο. Αλλά υπάρχουν πολλά επίπεδα τα οποία ουσιαστικά μας κάνουν 100% εξάρτητους. Το πρώτο είναι ότι απλώς παρέχουμε γνωμοδότηση και από εκεί και πέρα η αδειοδότηση είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί δεν δίνουμε άδεια. Ε, παρέχουμε γνωμοδότηση. Μπορεί να αμφισβητηθεί και έχει υπάρξει αμφισβήτηση κάποιε φορέ και ορισμένε φορέ μα έχει σταλεί και πάλι για επανεξέταση. Εμεί λοιπόν δεν δίνουμε καμία άδεια. Απλώ γνωμοδοτούμε. Υπάρχουν και πολλά άλλα επίπεδα. Το άλλο επίπεδο είναι ότι ο κλάδος πληρώνει προκαταβολή ουσιαστικά πληρώνουν για τη γνωμοδότηση και όχι για το αποτέλεσμα. Πληρώνουν τον ε, οργανισμό και ο οργανισμός μετά ορίζει εισηγητή και συνεισηγητή από κράτος μέλος για να αναλάβει το θέμα και ε, θα πληρωθούν εν ευθέτω χρόνο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Δεν δεσμεύονται δηλαδή για κάποιο αποτέλεσμα. Άρα τα χρήματα διατηρούνται για ένα άλλο επίπεδο. Ο εισηγητής και ο συνεισηγητής συναντιούνται για πρώτη φορά μετά από 120 μέρες εξέτασης και πολλές φορές διαφωνούν και αυτές οι διαφωνίες ε, ε συζητούνται μετά στην Ολομέλεια, στις οποία, στην οποία πρέπει να υπάρχει έγκριση με ειδική πλειοψηφία. Ο οργανισμός λοιπόν απλώς παρέχει δυνατότητες για ε, αυτά επιστημονικά στοιχεία, ε, κάνουμε αξιολόγηση ομολόγων, μπορούμε να δούμε τη διαδικασία γνωμοδότησης, αλλά δεν παρεμβαίνουμε στη διαδικασία λήψης απόφασης. Άρα είμαστε πλήρως ανεξάρτητοι. Η καινοτομία και τα τέλη αυτά δεν έχουν άμεση σχέση. Τα καινοτόμα φάρμακα εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο πλέον. Τα τελευταία 4-5 χρόνια άλλαξαν τα πράγματα και έχουμε ρηξικέλευτες καινοτομίες, γονιδιακές θεραπείες, κυταρικές θεραπείες, οι οποίες ε, είναι πλέον στην πρώτη γραμμή 25 για την επόμενη διετία. Και αυτά είναι κάτι τελείως καινούργια και τελείως καινοτόμα πράγματα η μεγάλη πρόκληση είναι να μην υπάρχει καινοτομία και τώρα η τεχνολογία και οι επιστήμη προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα με αλματώδη βήματα. Το πρόβλημα είναι η πρόσβαση και θα επανέλθω όταν θα συζητήσουμε για τον καρκίνο και τη βελτίωση για τα θέματα αυτά. Τώρα, το GDPR και η ερώτηση γι' αυτό. Η νομοθεσία αυτή θα μας ε, οδηγήσει πολλά καλά πράγματα θα μας δώσει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τη βάση δεδομένων Η ουσία ήταν να προστατεύσουμε τους ασθενείς, ε, τον κόσμο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους μεγάλους οργανισμούς που πουλούν τα δεδομένα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για επαναξιολόγηση της απόφασης και μπορούν να αποτελέσουν και ε, τα δομικά στοιχεία για επιπλέον έρευνα για πρόοδο της επιστήμης. Φυσικά, ανωνυμοποιούνται και φροντίζουμε να μην μπορεί κάποιος να εντοπίσει την αρχική πηγή, αλλά φυσικά αυτό δεν είναι δεδομένο 100%. πολλοί επενδυτές ε, δεν ε, ε, δίνουν στοιχεία τώρα με τόση προθυμία και φυσικά πρέπει να δούμε και τα δικά μας τα στοιχεία για να αξιολογήσουμε την αποφάση μας για το μέλλον. Μας υποστηρίζει βεβαίως η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ και Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις, κυρίως εκτός Ευρώπης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ανάγκη για κάποιες διευκρινήσεις ή αν θα αρκούν αυτές οι διευκρινήσεις ή θα πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση. Ε, είναι νωρί ακόμα για να το πούμε. Παρακολουθούμε την κατάσταση στενά και μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Τώρα, δύο λόγια για τον καρκίνο. Ξέρω ότι καθυστερώ. Η προτεραιότητα του καρκίνου είναι ευπρόσδεκτη. Όπως ε, είπα, η ευκαιρία να έχουμε για τους περισσότερους καρκίνους ε, τελική ε, θεραπεία είναι πρώτον πυλών, η επόμενη πενταετία, δεκαετία. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι η πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες, γιατί οι θεραπείες αυτές προϋποθέτουν όχι μόνο υψηλή τιμή και υψηλό κόστος, αλλά και πλήρη αναθεώρηση των συστημάτων υγείας ένα πρόσφατο παράδειγμα νοσοθεραπείας για τον καρκίνο. Υπάρχει μια πλήρης ακολουθία εμπειρογνωμοσύνης ε, και η παρασκευή των φαρμάκων ε, θα γίνει με διαφορετικό τρόπο και αυτό θα αλλάξει τελείως τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε επιθεωρήσεις, ε, την ποιότητα, το λεγόμενο GMP, τη διαδικασία διορδότηση. Κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να περάσουμε σε ένα χώρο που θα ε, γίνεται έγκριση σε κάποιες ε, πλατφόρμες που είναι ανταγωνιστικέ και να εγκρίνεται το τελευταίο σκέλος. Η πρόκληση λοιπόν του καρκίνου προϋποθέτει πολύ έντονες δραστηριότητες αναθεώρησης των διαδικασιών μας, ε, αλλά ε, είμαστε έτοιμοι από πλευράς ε, θεωρητικής, από, το, από πλευράς εργατικού δυναμικού όχι ακόμα, αλλά είναι πολύ καλό το γεγονός ότι αυτό το τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα είναι τόσο σαφές, διότι αφορά, αφορά πολλούς παράγοντες και σίγουρα ο οργανισμός φαρμάκων θα ε, παρέχει την τεχνική, επιστημονική και ε, πρακτική εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να πετύχει. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε και περνάμε στο τελευταίο τμήμα σήμερα το πρωί πριν από το κοκτέιλ που θα έχουμε. Θα συζητήσουμε με την Διεύθυνση Ανάλυσης και Ελέγχου τροφίμων και κτηνιατρικών προϊόντων. Δεν είναι ακριβώς ένας οργανισμός, αλλά νομίζω ότι έχει σχέση με τα υπόλοιπα που έχουμε συζητήσει σήμερα το πρωί. Οπότε, θα δώσω το λόγο στην Πάολα Κολόμπου. 7 με 10 λεπτά παρακαλώ. Και μετά φυσικά ε, στον Ευρωβουλευτή επαφή. Ευχαριστώ πολύ. Θα συντομέψω πάρα πολύ την παρουσίασή μου, να ξέρετε. Όπως είπατε, είμαστε μια διεύθυνση για την υγεία και την ασφάλεια. Είμαστε στην Ιρλανδική επαρχία και αποστολή μας είναι ο έλεγχος και η ανάλυση της εφαρμογής και υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τόσο στις χώρες ε, μέλη όσο και σε τρίτες χώρες. Και πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, δεν είμαστε ένας οργανισμός, αλλά κανονικά θα έπρεπε να είμαστε οργανισμός. Δηλαδή δημιουργηθήκαμε μετά την κρίση της ποκόδουσης κεφαλοπάθειας των βοηδών και γίναμε μια ανεξάρτητη υπηρεσία που έκανε ελέγχου σε διάφορες χώρες. Η αλλαγή έγινε τελευταία στιγμή από το Συμβούλιο και δεν γίναμε τελικά οργανισμός. Πάντως εδώ βλέπετε ότι ξεκινήσαμε με την ασφάλεια στην νομοθεσία, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε επεκτείνει τους οριζοντές μας και εξετάζουμε και την βιολογική γεωργία, ε, με την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, ε, κοιτάμε ιατρικά μηχανήματα, την ηλεκτρονική υγεία, άλλες δοκιμές και επεκτηνόμαστε όλο και περισσότερο. Είμαστε μόνο 165 προσωπικό οι 90 είναι ελεγκτές. Γιατί έχουμε και δραστηριότητες που δεν είναι ελεγκτικού χαρακτήρα. Και κάθε χρόνο προβαίνουμε σε 230 ελέγχους. Το 1 τρίτο αυτών είναι σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκθέσεις και τα σχόλια του ελεκτικού σώματος δημοσιεύονται όλα στην ιστοσελίδα μας. μόνο τα περιατρικών μηχανημάτων δεν δημοσιεύονται για την προστασία δεδομένων. Λοιπόν, σας είπα, κάνουμε τους ελέγχους, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι επίσης έχουμε και ελεγκτικά συστήματα που εξετάζουμε. Εξετάζουμε δηλαδή τα ελεγκτικά συστήματα των χωρών μελών και τρίτων χωρών για να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικά και κατά πόσο χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά στους ελέγχους μας, για τους ελέγχους μας, επισκευόμαστε διάφορα, μπορεί να είναι σφαγεία, μπορεί να είναι εργαστήρια, για να επιθεωρήσουμε και να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκεί είναι ικανοποιητικοί. Είναι σημαντικό λοιπόν να αντιληφθούμε ότι δεν επιθεωρούμε με μονομένες μονάδες, πρώτα απ' όλα γιατί είναι χιλιάδες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες, και καταλαβαίνω ότι είναι αδύνατον με 90 ελεγκτέ να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και έτσι καλλιώς δεν είναι καν στην εντολή μας. Ο κανονισμός μας μας ζητάει να κάνουμε συστημικούς ελέγχους. Προβαίνουμε σε συστάσεις και ζητούμε από τις ελεγκτικές μονάδες να προτείνουν ένα πρόγραμμα δράσης για να συμμορφωθούν στις συστάσεις μας και παρακολουθούμε μετά για να βεβαιωθούμε ότι όντως αυτό γίνεται. Κάποια νούμερα εδώ. Τα τελευταία χρόνια εκπονήσαμε 9.134 συστάσεις. Οι περισσότερες έχουν κλείσει, κάποιες παραμένουν σε κρεμότητα. Και όταν έχουμε έναν έλεγχο που είναι ιδιαίτερα προβληματικός, επιστρέφουμε για να επαληθεύσουμε κατά πόσο οι δεσμεύσει των αρμόδιων αρχών για να προβεί σε κάποιες διορθώσεις όντω υλοποιούνται ή όχι. Και έχουμε διαπιστώσει ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βεβαιωθούμε ότι οι συστάσεις μας ε, ακολουθούνται. Εδώ βλέπετε το ελεκτικό μας γαλαξία που είναι πολύ πλούσιος όπως βλέπετε. Στην αρχή είχαμε πιο λίγα πράγματα, τώρα έχουμε υγεία, τρόφιμα, ε, προστασία των ζώων, ε, για των φυτών, ζωοτροφές. Τώρα επικεντρώμαστε περισσότερο και στα ε, ιατρικά μηχανήματα, τις κλινικές δοκιμές, θα έχουμε μια αποστολή του χρόνου και ελέγχουμε επίσης και τις δραστικές ουσίες φαρμάκων που εισάγονται από άλλες χώρες στην Ευρώπη και ασχολούμαστε επίσης και με τη διαδικασία αμοιβές αναγνώρισης. Δυστυχώς όχι με την Κίνα και την Ινδία. Η δυσκολία που έχουμε είναι να συνεχίσουμε να καλύπτουμε όλα αυτά τα καθήκοντα με τους ίδιους ή και λιγότερους πόρους. Το ελεγκτικό μας πρόγραμμα για το 2020 βλέπετε ότι οι περισσότερες ε, έρευνές μας έχουν να κάνουν με την ασφάλεια τροφίμων, αλλά και με την υγεία που κερδίζει έδαφος συνεχώς. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το επόμενο πρόγραμμα εργασίας μας για το 2021 θα είναι για πρώτη φορά υπό έγκριση επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ βλέπετε πού βρίσκονται οι συναδελφοί μας, πού πήγανε τον Οκτώβριο μάλλον, και στην Ευρώπη αλλά και ανά τον κόσμο. Θέλω να ολοκληρώσω τονίζοντας κάποιες ιδιαίτερες δραστηριότητές μας όπου δραστηριοποιηθήκαμε πολύ τα τελευταία χρόνια, είναι η προστασία των ζώων. Έχουμε ελέγχους στις δύο προτεραιότητές μας που είναι οι μεγάλες ε, μονάδες εκμετάλλευσης και οι μεταφορές. Για τις μεταφορές έχω καλά νέα γιατί σε 18 χώρες μέλη την τελευταία χρονιά ελέγξαμε για τις μεταφορές που γίνονται το καλοκαίρι και διαπιστώσαμε ότι χάρη στην ε, δικιά μας προσπάθεια να πείσουμε τις χώρες μέλη να αναλάβουν δράση, ότι βελτιώθηκαν τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων, είναι μια ευθύνη της πολιτικής, έτσι. Εμείς κάνουμε εκθέσεις και αξιολογώντας τα εθνικά προγράμματα δράσης. Και όπως είπα και νωρίτερα, είμαστε και υπεύθυνοι για την δημιουργία εναρμονισμένων δικτών προκειμένου να μπορούμε να δούμε ο κίνδυνος που έχει να κάνει με τα φυτοφάρμακα μειώνεται τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχομαι στην τελευταία διαφάνεια που ήθελα να σας δείξω είναι για τα ιατρικά μηχανήματα. Έχουμε ήδη κοινή αξιολόγηση με τον προηγούμενο κανονισμό που οδηγεί σε μια μείωση των ε, οργάνων που πιστοποιούν, αλλά και όσον αφορά το εύρος. Και έτσι το αποτέλεσμα είναι ότι τα ιατρικά μηχανήματα είναι περισσότερο ασφαλή από ό,τι κατά το παρελθόν. Επίσης, κοιτάζουμε και τις νέες εφαρμογές. Ε, περιμένουμε 20 πιστοποιημένους οργανισμούς το, να έχουμε τον Ιανουάριο και λειτουργούμε πλήρως. Περιμένουμε τις ε, αιτήσει λοιπόν από τα όργανα που κοινοποιούν. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είχατε 10 λεπτά στη διάθεσή σας, δεν τα αξιοποιήσατε όλα, οπότε θα σας δώσουμε πίστοση ένα λεπτό κάτι την επόμενη. Καταρχήν λοιπόν ο Κονιατσικά έχει τώρα το λόγο. Ακούσαμε μόλις τώρα ε, μια παρουσίαση όπου υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριότητα για αυτήν την ε, ε, μονάδα. Οπότε η τελευταία διαφάνεια που είδαμε εδώ, η μία από τι τελευταίε διαφάνειε, ε, είναι πλέον σημαντική. Δηλαδή, το νέο πρόγραμμα εργασιών τη Επιτροπή σε ό,τι ειδικότερα αφορά το ζήτημα τη μικροβιακή αντοχή. Γνωρίζω πω είναι ένα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα. Προβαίνεται και σε ελέγχου σε σχέση με αυτό το θέμα. Και θα θέλαμε πολύ να έχουμε κάποια στιγμή την ευκαιρία να ακούσουμε μία εις βάθος ανάλυση από την πλευρά σας σε ό,τι αφορά το ανάλογο θέμα. και συχνά αναφερόμαστε ε, σε αυτήν την ε, γενική διεύθυνση χωρί όμω να αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώ κάνει. Μιλάμε για επιβολή τη νομοθεσία, τη ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, των ζώων τροφών, ε, την υγεία των ζώων και ούτω καθεξής. Χωρί να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι η κυρίω αρμόδια γενική διεύθυνση. λοιπόν όταν ε, ε, οι γνωμοδοτήσει από την πλευρά αυτή τη Γενική Διευθύνση δεν θα πρέπει να αξιοποιούνται μόνο από την Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να αξιοποιούνται και από εμά, από το Κοινοβούλιο, κατά την προετοιμασία των δικών μα εκθέσεων, ψηφισμάτων κ.ο.κ. Θα ήθελα να, να θέσω ένα ερώτημα. Ε, ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία αποφασίζεται ποιοι θα είναι οι επόμενοι έλεγχοι που θα δεξάγεται. Αυτά από την πλευρά μου και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχίσουμε μια πολύ ενεργή ενεργό συνεργασία ανάμεσά μας γιατί ε, θα είναι πολύ χρήσιμη και για όλα τα μελλοντικά θέματα που θα εξετάσουμε εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η κυρία Σπυριακτώρα τώρα από, το, από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε παρακολούθησα πολύ προσεκτικά το πρόγραμμα εργασιών για το 2019 αυτής της Μονάδας Ελέγχων και Αναλύσεων ε, και εγώ από την πλευρά μου υποστηρίζω ιδιαίτερα την δίαιτα vegan, οπότε θα μπορούσαμε να αποφύγουμε βέβαια πολύ μεγάλο κομμάτι όλων αυτών των εργασιών εάν δεν είχαμε ζώα τα οποία προορίζονταν για να κατανάλωση. Πάντως μας είπατε ότι το 2021 για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει ε, το σχέδιο για τους ελέγχους. Γιατί λοιπόν αυτό δεν συνέβαινε μέχρι τώρα μια τέτοια έγκριση. Ευχαριστώ. Κυρία Ζανκάμπ τώρα για το Ιγκούα. Θα μιλήσω Ολλανδικά, κυρία Κολόμπο. Είμαι από το κόμμα για την προστασία των ζώων, με τον συνάδελφο. Θέλουμε περισσότερη προστασία των ζώων και χαίρομαι που εσείς δίνετε σημασία σε αυτό το θέμα. Πηγαίνετε στα σφαγεία, ασχολείστε με τη μεταφορά των ζώων κτλ. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν για τους ελέγχους και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ανάμεσα στην Ουρουάη και την Αργεντίνη μεταφορά. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκεί και για την υγεία των ανθρώπων, διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει ντόπινγκ εκεί με τα φάρμακα που δίνουν στα ζώα. Λοιπόν, έγιναν κάποιοι έλεγχοι και φάνηκε ότι μετακινούνται, μεταφέρονται τα ζώα με τρόπο που κινδυνεύει τελικά ο κόσμος, χωρίς δηλαδή να υπάρχει προστασία. Και όμως, τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν προσφέρονται τα ζώα. Δεν προστατεύονται. Δεν θα ήταν καλύτερα λοιπόν οι έλεγχοι που γίνονται να μην ανακοινώνονται προηγουμένως, γιατί όταν ανακοινώνονται παίρνουν τα μέτρα τους οι άνθρωποι που κάνουν τις μεταφορές. Και για την περίπτωση αυτή Ουρουγουάη και Αργεντινής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε τη το δικό σα το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγέ από εκεί δεν τηρούν τους ε, κανόνες πλήρω. Οπότε ρωτάω, αυτό δεν πρέπει να το πάρουν πάρα πολύ στα σοβαρά και συμβαίνει συχνά οι δικοί σας οι έλεγχοι να μην λαμβάνονται υπόψη, να αμφισβητούνται τελικά τα συμπεράσματα από αυτούς. Thank you. Any other Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο άλλο ε, συνάδελφο που θέλει να θέσει ερωτήματα. Εάν όχι, μπορείτε να απαντήσετε στα όσα επόθηκαν μόλι τώρα και να προσθέσετε και περαιτέρω θέματα αν θέλετε. Ναι, ευχαριστώ πρώτα. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή αντοχή. Ήδη έχουμε προβεί σε δύο σειρέ μόνο σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, σωστή, τη δέουσα χρήση ε, τον φαρμάκων σε ό,τι αφορά τη μικροβία αντοχή ε, σε σχέση με βακτήρια και σε σχέση με ζώα και από την συνάδελφο εδώ από το ECDC προβαίνουμε σε ελέγχους One Health, δηλαδή ενιαία προσέγγιση για την υγεία. Δηλαδή, προσπαθούμε να έχουμε κοινή εξέταση σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, την κτηνιατρική χρήση και τι περιβαλλοντικέ επιπτώσει αλλά ε, δυστυχώ αυτό θα, το, μπορούμε να το κάνουμε μόνο με κατόπιν ετήματο, κατόπιν πρόσκληση, Δεν μπορούμε να αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να το κάνουμε από μόνοι μα, αλλά αποτελεί πραγματικά αυτό ένα νέο τρόπο για να εξετάζουμε ένα πρόβλημα και συγκεκριμένα αυτό της μικροβιακή αντοχής. Δεν μπορούμε δηλαδή ε, αποσπασματικά ο καθένα από την πρέπει να το ε, προσεγγίζουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια με βάση τα οποία ορίζουμε το πρόγραμμα εργασιών μα, καταρχήν έχουμε ένα, μια βασική σειρά, δηλαδή ότι λέμε κατά συγκεκριμένη περίοδο ετών θα πρέπει να εξετάσουμε ένα συγκεκριμένο κράτο μέλο σε ό,τι αφορά συγκεκριμένου τομεί και από εκεί μετά υπάρχουν κάποιε έκτακτε περιπτώσει, στο πλαίσιο δηλαδή των οποίων το σύστημα συλλογή πληροφοριών μα μας καταδεικνύει, αυτό το σύστημα RAPS, καταδεικνύει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει ανακύψει. Για παράδειγμα, εμφάνιση σαλμονέλα, ε, μια συγκεκριμένη, συγκεκριμένη τροφίμων. Εκεί λοιπόν δίνουμε προτεραιότητα στο λόγο ζήτημα. Και εστιάζουμε σε πολύ συγκεκριμένους ε, τομείς που μας ενδιαφέρουν, για παράδειγμα όπως η ευημερία των ζώων, και αποφασίζουμε δηλαδή να θέσουμε ένα τέτοιο τομέα σε προτεραιότητα για το πρόγραμμα εργασιών και εστιάζουμε εκεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι τρίτε χώρε, υπάρχουν και αιτήματα πρόσβαση στην αγορά. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες, τρίτε χώρε, οι οποίε ζητούν να προβούν σε εξαγωγέ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο συγκαταλέγουμε ελέγχου σε αυτέ τι δύο χώρε στο πρόγραμμα εργασιών μα. Σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο τώρα ελέγχων, αυτό το πρόγραμμα ελέγχων, αυτό αναπτύσσεται από κοινού και με τα κράτη-μέλη και ο νέο οικονομισμό ε, για τι επισημέ διατάξει που τώρα πρόσφατα, ή μάλλον τώρα σε λίγο θα αρχίσει να ε, ισχύει, στις 14 δηλαδή Δεκεμβρίου, προβλέπει ακριβώς ε, επίσημη έγκριση από την πλευρά της Επιτροπής του Ανλόγου προγράμματος ελέγχων. Αυτό είναι ο μόνος λόγος. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το ζήτημα των λέγων, έχουμε ιδιαίτερα εστιάσει στο κρέα αλόγων. Όχι μόνο σε τρίτε χώρε, αλλά και εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή προβλέπουμε σε μια σειρά δοκιμών, ακριβώ σε σχέση με αυτό το θέμα του κρέατο αλόγου, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο υπάρχουν ακόμα ε, φαινόμενα απάτη σε αυτό το τομέα. Και ε, σύντομα θα έχουμε και τα αποτελέσματα από αυτέ τι σειρέ δοκιμών. Εξετάζουμε όμω, όπω σα είπα, και το ζήτημα του αλλογή του και σε τρίτε χώρε. Και έχετε ε, δίκιο σε αυτό που είπατε, ότι δηλαδή ε, μα ενόχλησε ιδιαίτερα το γεγονό ότι σε τρίτε χώρε, όταν μεταβαίναμε εκεί για να κάνουμε τον έλεγχο, όταν φτάναμε σε αυτόν τον στάβλο, ε, όπου υποτίθεται πω βρίσκονταν τα, τα ζώα, ε, δεν υπήρχε ζώο και ήταν πεντακάθαρη εν λόγω ε, Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι προσπαθούσαν κάτι να κρύψουν από την πλευρά του αυτέ τι τρίτε χώρε. Όμω αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να προβούμε σε ευνίδιε επισκέψει. Χωρί δηλαδή να, ε, να υπάρξει προειδοποίηση. Μπορούμε να καταφτάσουμε σε μια τρίτη χώρα και να πούμε αύριο θέλουμε να μεταβούμε στην λόγω εγκατάσταση. Και ενώ σε κάποιε περιπτώσει αυτό είναι δυνατό και μπορούμε να το ζητήσουμε, στη Λατινική Αμερική, στι χώρε δηλαδή τη Λατινική Αμερική, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Δεν μα το επιτρέπουν. Και επίση υπάρχει βέβαια και το ζήτημα τη διαφορετική νομοθεσία που ισχύει εδώ, αφενό στι δικέ μα χώρε και στι τρίτε χώρε αφετέρου. Ειδικότερα δηλαδή σε ό,τι αφορά τα επίπεδα, τα, ε, ε, ε τα υπολείμματα, επίπεδα δηλαδή ε, υπολείμματων συγκεκριμένων ουσιών και ούτω καθεξής. Δηλαδή, εκεί είναι δυνατόν να γίνει η σφαγή αλόγων για κατανάλωση του κρέατος εφόσον δεν, έχουν, ε, δεν έχει υποβληθεί το σχετικό ζώο σε κάποια θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή δηλαδή, κατά του τελευταίους έξι μήνες. Κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό. Τώρα υπάρχει για παράδειγμα περίπτωση της Βραζιλίας της Ταϊλάνδης για τις οποίες χώρες με βάση τα αποτελέσματά μας προβαίνουμε στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Ειδικότερα δηλαδή όταν υπάρχουν ε, συμφωνίες εμπορίου ή διαπραγματεύσεις για τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα πιο πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το, τη, τη, τη, τη, συμφωνία με την Μερκοσούρ, αυτό είναι ένα ολόκληρο καινούριο ζήτημα που θα μπορούσαμε να συζητούμε για μία ώρα, για να μην αναφερθώ καν στο Brexit. Όλα αυτά δηλαδή θα άρχισαν περαιτέρω συζήτηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε εδώ λοιπόν με την πρωινή μα συνεδρίαση και θα περάσουμε τώρα στο κοκτέιλ. Εδώ σε αυτή την αίθουσα θα λάβει χώρα και θα έρθει, δηλαδή θα έρθω σε λίγο τα φώτα. Ευχαριστώ πολύ.